Okay, dear members, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο στην ημερήσια διάταξη και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας για την ανταλλαγή απόψεων τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά Κατάινεν, που εντέλεσε και Πρωθυπουργό ε, της Φιλανδίας από το 2011 μέχρι το 2014, δεν κάνω λάθος, και τώρα είναι αντιπρόεδρος ε, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Ένας άλλος επίτιμος καλεσμένος μας ε, είναι ο κύριος Βίλχελμ Μόλτερερ, πρώην βουλευτής της Αυστριακής Βουλής και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τάπαζας Επενδύσεων από το 2011. Έχει ειδική αρμοδιότητα την πολιτική συνοχή. Σήμερα το πρωί εγκρίναμε την ε, γνωμοδότησή μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωμοδότηση προς την, έκθεση, την κοινή έκθεση των Επιτροπών Οικονομίας και προϋπολογισμών. Μετά τις ψηφοφορίες που θα γίνουν τον Απρίλιο στις αρμόδιες επιτροπές θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη θέση και στόχος της δικής μας επιτροπής είναι να εξασφαλίσει μία συμπληρωματική σχέση μεταξύ του νέου Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της νέας γενιάς ε, της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ε, να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να αξιοποιήσουν αυτό το νέο ταμείο και εν ώψη της αναθεώρησης της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 όλα αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα έλεγα να ακολουθήσουμε την ε, γνωστή μας διαδικασία, να δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για μια σύντομη παρουσίαση για το τρέχον και μέλλον έργων τους και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους συντονιστές για ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά στους υπόλοιπους βουλευτές. Και οι δύο καλεσμένοι μας είναι πολύ άσχολοι, γι' αυτό και μέχρι τις 4 και 4 θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα γιατί δεν ε, δίνονται να παραμείνουν περαιτέρω οι καλεσμένοι μας. Γι' αυτό θα σας θέλουμε παρακαλούσα να υποβάλλετε συναπτικά τις ερωτήσεις σας, ώστε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας στο έπακρο. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γύρκη να Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτήν την πολύ σημαντική επιτροπή. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός για να αφήσουμε χρόνο για τη συζήτηση, να ακούσω τις απορίες σας, ε, τα σχόλιά σας και να απαντήσω. Δεν θα σας κάνω διάλεξη. Το βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ότι θα επιφέρει προστιθέμενη αξία. Η προσθετικότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, κάνει θαυμάσια δουλειά ε, δανείζοντας 60 με 70 δισεκατομμύρια το χρόνο για επενδυτικά προγράμματα και το νέο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα συμπληρώσει το έργο της ΕΤΕΠ και θα επικεντρωθεί σε πιο υψηλού κινδύνου σχέδια. Και εδώ έχουμε δύο πτυχές. Η μία πτυχή αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έκανα μία περιοδία, μέχρι στιγμής έχω επισκεφτεί 10 χώρες, απομένουν άλλες 14 ε, που θα επισκεφτώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Και ένα πολύ κοινό σχόλιο που ακούω το άκουσα και στη Γερμανία και τη Δευτέρα στην Κύπρο, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετό μετοχικό κεφάλαιο. Σε πολλέ χώρες έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή όμω δεν έχουν μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορούν να ζητήσουν στι αγορέ κεφάλαια. Και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάμε και με το Ταμείο το Επενδυτικό. Δεν θέλουμε εμείς να υποκαταστήσουμε τις τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, απλώς θα γεφυρώσουμε ένα χάσμα που υπάρχει, το χρηματοδοτικό χάσμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε σχέδια υποδομών, το Ταμείο θα πρέπει να επιλέξει σχέδια που δεν θα μπορούσαν να δουν το φως της ημέρας χωρίς αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο του επιμερισμού του κινδύνου που το χορηγεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η προσθετικότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία ως ε, συγχρηματοδοτικό στοιχείο για ε, σχέδια που θα, θα δώσει εγγύηση στο ΕΦΣΙ, το Ταμείο έτσι δηλαδή οι ιδιότητες επενδυτές ε, θα επενδύουν τα χρήματά τους και εμείς ε, θα προσθέσουμε κάποια στοιχεία επιμερισμού του κινδύνου και υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότηση και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτός ο συνδυασμός ε, είναι εφικτός και να απόκειται στα κράτη-μέλη να τον αξιοποιήσουν. Ένα επιπλέον στοιχείο της επενδυτικής πολιτικής, πολύ σημαντικό, είναι η ανεξαρτησία της επιλογής, της διαδικασίας επιλογής των σχεδίων. Να μην υπάρχει πολιτική επίδραση στην επιλογή των σχεδίων. Να Είναι αποπολιτικοποιημένη διαδικασία. Στις επισκέψεις μου στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερες συναντήσεις με επενδυτές ε, του ιδιωτικού τομέα, η ερώτηση που ακούω συχνά είναι ποιος θα επιλέξει τα, τα σχέδια. Και τους διαβεβαιώ ότι θα είναι μια ανεξάρτητη επενδυτική επιτροπή και ο διορισμός των μελών της ε, θα γίνει από ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες, ε, θα εξετάζουν τα σχέδια και θα δίνουν το πράσινο φως για τις εγγύσεις. Δεν θα είναι πολιτικού χαρακτήρα η επιλογή, ούτε θα υπάρχει γεωγραφική υποχρεωτική κατανομή ή τομεακή υποχρεωτική κατανομή. οι εμπειρογνώμονες ε, της, ε, τράπεζας, ε, της Επιτροπής Επενδύσεων με αξιοκρατικά και μόνο στοιχεία θα επιλέγουν τα προγράμματα, τα σχέδια προς επένδυση. Αν δεν εξασφαλίσουν αυτή την εξαρτησία θα πάει στράφη όλο το ταμείο. Επίσης μας ρωτάνε οι επενδυτές από πού θα προέλθουν τα κονδύλια, από ποιες δημοσιονομικές γραμμές, από πού θα προέλθουν οι ευρωπαϊκές εγγύσεις. Οι επενδυτές θα θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις πηγές αυτών των κονδυλίων και ε, ρωτούν ότι θα γίνουν ετήσιε διαπραγματεύσει στον προπολογισμό, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει τεράστια αβεβαιότητα. Εγώ είπα ότι η, προ... Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφέστατη. Ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ασαφεί ε, αιτήσει διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό, για να υπάρχει προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου και να γνωρίζουν οι επενδυτέ από πού και θα προέλθουν τα κονδύλια και ποιο θα είναι το ύψος τους. Επίσης, ε, δεν χρειάζεται, ε, όπως είπαμε, να δοθούν 16 δισεκατομμύρια επενδύσεις, λέει το Κοινοβούλιο. Θα σας εξηγήσω όμως, ο κύριος Μόλτερ, τι θα συμβεί αν δεν έχουμε αυτές τις εγγύσεις 16 δισεκατομμύριων. Ε, και θα δυσκολέψουμε την ΕΤΕΠ, αλλά και θα υπονομεύσουμε την πιστοληπτική ικανότητα και την αξιολόγηση της ε, επενδυτικής τράπεζας, τα 3α. Επίσης θα πρέπει το ταμείο να είναι αξιόπιστο, διαφανές, ε, σαφές, να τεθεί σε εφαρμογή γρήγορα και η διαδικασία επιλογής των σχεδίων να είναι ανεξάρτητη από και να γίνεται αμυγός με αξιοκρατικά κριτήρια. Έτσι θα έχουμε ένα λειτουργικό ταμείο που θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σχέδια κινδύνου υψηλού. Ακούστηκε γιατί, ακούστηκε πολλά γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσω να χρησιμοποιήσει ως πηγή χρηματοδότησης το ορίζον 2020 και το συνδέοντας στην Ευρώπη. Και υπάρχει ένα λόμπι πέρα της χρήσης των διαρθρωτικών κονδύλιων ή του το Γεωργικού Ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ριζικά αντίθετη με την πρόταση αυτή και ο λόγος που χρησιμοποιούμε το Horizon 2020 και το ΣΕΦ, το Μηχανισμό τη Διευκόλυνση μάλλον συνδέοντα στην Ευρώπη, είναι γιατί τα προγράμματα, τα σχέδια που χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι τα ίδια με αυτά που θα χρηματοδοτούσε και το συνδέοντα στην Ευρώπη ή Horizon 2020. Οπότε θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα χρησιμοποιήσουμε 2,7 δις για την έρευνα δίνοντας επιδοτήσεις ή αν θέλουμε ε, με μόχλευση να έχουμε δεκαπλάσιο ποσό από τα 2,7 δις και έτσι να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα με πολύ περισσότερα κονδύλια από 2,7 δις με τη χρήση χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Κοιτάξτε τις χώρες που έχουν υψηλό ποσοστό έρευνας και και ανάπτυξη σε σχέση με το ΕΠ Εκεί χρησιμοποιούνται πολλά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Φυσικά δίνονται και επιχορηγήσει, αλλά χρησιμοποιούνται και πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα. Ε, μόλις επέστρεψα από την Κύπρο και εκεί δύο πανεπιστήμια με ιδιαίτερη περηφάνεια παρουσίασαν τα σχέδιά τους που δανειοδοτήθηκαν από την ΕΤΕΠ. Και στην Γαλλία, το Πανεπιστήμιο Έξαν Μαρσέγ, με πολύ χαρά μας περιέγραψε την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μου είπαν ότι με το που θα τεθεί σε ισχύ το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Πανεπιστήμιο θα επωφεληθεί και από νέα κονδύλια, ε, ιδιαίτερα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα που θα επενδύσει σε σημαντικές υποδομές ερευνητικές. Αυτό για όσου φοβούνται ότι η βασική έρευνα δεν θα υποφεληθεί από το ΕΦΣΙ. Λάθο. Αυτό ήδη συμβαίνει και θα συμβεί και στο μέλλον. Βέβαια, η πλειοψηφία της ε, βασικής έρευνας ε, χρηματοδοτείται κυρίως από, ε, από δημόσια κονδύλια. Αλλά οι επενδύσεις για άλλα, άλλους τομείς της μπορούν να χρηματοδοτηθούν και έχουν και στο παρελθόν χρηματοδοτηθεί από χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Οπότε, το συνδέοντας την Ευρώπη και ορίζοντας το 2020 μαζί αντιπροσωπεύουν το 70% του τίτλου 1α. Και αν αυτοί οι πόροι χρησιμοποιηθούν θα αφορούν το βελαιό και το έρασμο. Αυτά δεν επωφελούνται από χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Αυτά και περιμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλια, τις συμβουλές σας και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις ώστε να συζητήσουμε και τώρα να δώσουμε τη σκητάλη στον κύριο Μόλτερ. Κύριος Μόλτερ, γεια σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' συγχαρητήρια που τα καταφέρατε όσον αφορά την ψηφοφορία για το ε, ζήτημα το οποίο συζητούμε. Μου θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογο αυτό και τελικά το θέμα είναι ανάπτυξη και <clears throat> απασχόληση. Για την αιτία αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή και χέρι χέρι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια έξτρα όθηση ε, στην ε, ανάπτυξη και την απασχόληση. Αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε πώς θα γεφυρώσουμε το χάσμα των ε, επενδύσεων, γιατί όπως ξέρετε ακόμα έχουμε 15% κάτω από το επίπεδο του 2007, 15% ενώ άλλοι, άλλοι και τα προηγούμενα χρόνια κάλυψαν το χαμένο έδαφο. Εμεί ακόμα ε, είμαστε ουραγοί, έχουμε καθυστερήσει. Αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτό το κενό το επενδυτικό. Υπάρχει και ένα άλλο αποτέλεσμα, δηλαδή πέφτουμε σε ανταγωνιστικότητα. Επομένω, εάν ενθαρρύνει κανεί τι επενδύσει, δεν ε, βελτιώνει την απασχόλησή του, αλλά επίση δίνει και μειώθηση στην Ευρώπη προ ένα καλύτερο επίπεδο ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά. Και είναι σημαντικό, επομένω, και τα δύο αυτά στοιχεία θα λάβουμε υπόψη να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και επίσης να βοηθήσουμε ανάπτυξη και απασχόληση και ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Και είναι αυτό πάρα πολύ βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας μας. Ακούσατε είπε ο Επίτροπος ε, Κατάινεν και σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επιμεδίσεων ε, υποστηρίζει και τις πολιτικές ανάγκες αλλά επίσης αναλαμβάνουμε δράση εάν ε, η αγορά δεν μπορέσει να βοηθήσει τα πράγματα και πώς είναι η κατάσταση στην αγορά όλοι ξέρουμε για αυτό το το κενό της, ε, ε, των επενδύσεων. Ξέρουμε ότι υπάρχει με την παραγωγικότητα στη δε αγορά. Τώρα έχουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση και σύμφωνα με την οποία ε, δεν έχουμε πρόβλημα πλέον της ρευστότητος και στον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα και στις τράπεζες. Το πρόβλημα όμως στην Ευρώπη εδώ είναι άλλο, ότι ακόμη οι εμπορικές τράπεζες δεν μπορούν να λάβουν σημαντικούς κινδύνους. δεν μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε μια κεφάλαια αγορά η οποία είναι οίκιστα ε, ανεπτυγμένη που είναι τόσο σημαντική και οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό κομμάτι από το πρόγραμμα Juncker είναι ότι θα πρέπει εντατικά να προβληματιστούμε πώς θα άρουμε αυτούς τους φραγμούς που εμποδίζουν τι επενδύσεις. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναφαντώνει υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Την υποστηρίζουμε και θεωρούμε ότι θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη έχει δραστηριοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πέρσι είσαμε 77 δις. 77 δις δανείσαμε στην Ένωση και Ω πρωτοβουλία έχουμε να υποστηρίξουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχείρησεις, τις ε, υποδομές, αποτελεσματική χρήση των πόρων και την καινοτομία. αυτέ είναι οι προτεραιότητες μας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί είναι ένα παραπάνω ε, εργαλείο τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πλωστάσιο από πλευρά ΕΤΕ και είναι και ποσοτική βελτίωση αλλά και ποιοτική. Επομένως, είναι ένα βασικό ζήτημα. Το EFSI για μας αποτελεί μια εγγύηση ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο πρώτα, να λάβουμε περισσότερο κινδύνους και νέες επιχειρήσεις και επίσης έχουμε τώρα μια καινούργια γενιά από χρηματοοικονομικά προϊόντα και σας υπεβιώνω αυτό το οποίο σας είπε ο Επίτροπος για μας πολύ σημαντικό είναι να είναι ισχυρή και να είναι ε, ικανής ε, ε, αρκετού βεληνικού σε αυτή η εγγύηση, να μπορεί να κινητοποιηθεί αμέσως, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια προϋπόθεση που εμείς τη, τη, θεωρούμε, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε αξιολόγηση τριπλού αλφα, αλφα, αλφα, αλφα, γιατί αυτό είναι ο πυρήνας της ε, τέμας τόσο ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις. Άρα ποιότητα της εγγύησης πρώτον, δεύτερον ζητούμε εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσετε μία ε, ισχνή δομή διευθυντική, χωρίς δηλαδή πολλά άτομα και αν ε, απευθυνθείτε στον κόσμο θα, θα, θα δείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον επένδυσης σε έργα και projects. Όμως χρειάζεται επαγγελματική διαδικασία επιλογής και χρειάζονται επαγγελματίε οι οποίοι να ασχολούνται με την ε, εγγύηση. Και αν πολιτικοποιήσει κανείς ε, όλα αυτά τα πράγματα τότε θα φέρει μόνο εμπόδια θα δυναμητήσει την όλη ιδέα. Γι' αυτό είμαι κατηγορηματικός. Κατά τρίτον, ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι η προσθετικότητα όπως συμφωνήσαμε με την ε, Κομισιόν. Γιατί έτσι έχουμε τα σωστά κίνητρα ούτω ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων το συντομότερο δυνατό. Σας είπε επίσης ο Επίτροπος για ε, τρία άλλα παράθυρα ευκαιρίας για παραπάνω υποστήριξη. Ε, ΜΜΕ σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων γιατί βλέπουμε ότι η αγορά ε, χρειάζεται στήριξη των ε, mid-caps, των μεσαίας κεφαλοποίησης εταιριών, οι οποίες δηλαδή ε, έχουν, είναι εξωστραφείς σε εξαγωγές και οι οποίες έχουν τώρα έχουν στριμωχτεί αρκετά όσον αφορά την χρηματοδότηση. Δεύτερο, δεύτερος τομέας είναι τι θα κάνουμε με την καινοτομία. Η παιδεία, η κατάρτιση, οι δεξιότητε, όλα αυτά για μας είναι θέματα κλειδιά για να μπορέσουμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα. Κατά τρίτο λόγο είναι η οι υποδομές. Και βέβαια λέμε για υποδομές με την ευρία έννοια. Όχι μόνο δηλαδή δρόμους και, και τρένα, αλλά και την κοινωνική υποδομή. μήμοι έξω επομένως, καινοτομία, υποδομές. Αλλά υπάρχει ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμούμε, δηλαδή η δυνατότητα παροχής συμβουλών. Ή το λέει και ο κανονισμό ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα τέτοιο κόμβο ε, συμβουλευτικό και να είναι κοινή πρωτοβουλία για να υποστηρίξουμε και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην προετοιμασία των projects, στην ε, προετοιμασία εφαρμογή του, παρακολούθησή του κλπ. Και αυτό ισχύει και με τα χρηματοοικονομικά ε, εργαλεία και επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία δυνατοτήτων όσον αφορά και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Επομένως, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και αυτός ο κόμβος της ε, παροχής συμβουλών. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες, ήδη κάποιες έχουν να τρέχουν, ας πούμε το κόμπας. Και θέλω να σας πω το τελευταίο ότι για μας η συνοχή είναι μια υψίστη προτεραιότητα. Από τότε που συγκροτηθήκαμε τότε που ε, αρχίσαμε να υπάρχουμε το 58 λοιπόν τότε για μας είναι ένα θέμα κλειδί πολιτικού χαρακτήρα το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων δεν θα υποκαταστήσει κάτι θα συμπληρώσει τα όσα ήδη υπάρχουν για την πολιτική συνοχή ο δανεισμός έφτασε το 30% όσον αφορά την συνοχή. Μιλάμε για 25-30 δις. Και αυτό το οποίο θα καταφέρουμε την γεννή πρωτοβουλία είναι το εξής. Θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των υπαρχών των εργαλείων μας όσον αφορά την συνοχή. Γιατί αν δείτε τα πράγματα μακροπρόθεσμα, η μόχλευση και η αξιοποίηση του δημόσιου κορβανά για τι ανάγκε που υπάρχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό και για μα το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι μια αφιτηρία πάρα πολύ σημαντική ούτω ώστε να υποστήριξουμε την πολιτική συνοχή μακροπρόθεσμα. Τι να πω άλλο για να σας πείσω. Για μας επομένως είναι αυτό, αυτή η προετοιμασία, η, η προτεραιότητα, η συνοχή. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της πολιτικής της συνοχής με το καινούριο ΕΦΣΥ. Και αυτό θα ωφελήσει και τα 28 κρατη Δεν έχουν τίποτα ποσοστώσεις. Θα ε, συνοηθούμε με εθνικούς φορείς, με περιφερειακές ενώσεις και φορείς και γι' αυτό και νομίζω ότι θα δοθεί μια έξτρα όθηση. Και γι' αυτό σας ζητώ, συνάδελφοι, εδώ στο Κοινοβούλιο να μπορέσετε να ε, κάνετε κι εσείς ό,τι μπορείτε για να λάβει σάρκα και ωστά το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και το χρειάζεται η Τράπεζα Επενδύσεων, το χρειάζεται η Ευρώπη ούτως ώστε να υπάρχει ανάπτυξη και επενδύσεις. Ευχαριστούμε, λέει ο, η πρόεδρος προς τον κύριο Μόλτερ. Και τώρα. Θα ξεκινήσουν οι συντονιστές και κατόπιν τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Α, για το ΕΛΚΟ, κύριο Φανίστελο. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε και τους δύο εδώ και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχετε ευρείτε το χαρτοφυλάκιο, κύριε Κατάινεν, κύριε Αντιπρόεδρε. Και κρατάτε αυτή την καλή συνήθεια να, για τακτική ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα, για πολλά διάφορα και πολλά και διάφορα θέματα των ε, δραστηριοτήτων σας. Σήμερα είναι η μέρα του ΕΦΣΥ. Βέβαια το πρωί είχαμε εκτενή ψηφοφορία και συζήτηση, τώρα είναι το after party ουσιαστικά με εσά. Ε, δεν πρόκειται να μας πείσετε για τα πάντα. Μετά από δύο μήνε ίσως ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις όχι μόνο με εσά, αλλά και με το Συμβούλιο φαντάζομαι. Το θεμελιώδες ζήτημα είναι ότι ήδη στον κανονισμό μας είχαμε πολλούς μηχανισμούς που ε, αφορούσαν τα περιστρεφόμενα κονδύλια, ακόμη και το χρηματοπιστωτικό των ε, ε, χρηματοπιστωτικό μας κανονισμό τον αλλάξαμε για να επιτρέψουμε τέτοιες μεθόδους. Επίσης ε, είχαμε και το ορίζον 2020 με τη δυνατότητα επιμερισμού του κινδύνου. Οπότε δεν είναι καινούργια όλα αυτά τα στοιχεία. Ίσως η ένταση τους και η συγκέντρωση είναι το καινούργιο στοιχείο. Εγώ θα ήθελα πάντως ε, και με τους δυο σας και μεταγενέστερη συζήτηση για να ενημερωθούμε για τα επιχειρησιακά προγράμματα, για τα συμβόλαια εταιρικής σχέσης ε, με βάση τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Γιατί τα εργαλεία υπάρχουν. Τα αξιοποιούμε όμως, γιατί υπάρχει ο μηχανισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τον ε, εκμεταλλευόμαστε. Είμαστε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά πλευρά του Συμβουλίου είναι κάπως απρόθυμη, ενώ υπάρχει δυνατότητα. Και είναι και η στιγμή να δούμε πώς θα μάθουμε πολλά πράγματα, τι θα διδαχθούμε από τη νέα πρωτοβουλία. Και τη χρήση των άλλων εργαλείων τα οποία δεν θα πρέπει να αλληλοαποκλείονται. Θα πρέπει τα επιτελεία σας ε, να συνεργάζονται με τις ήδη φυστάμενες αρχές διαχείρισης. Να μην υπάρχει αντιπαλότητα, είναι πολύ σημαντικό. Και είπαμε το πρωί ότι θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει την κατάσταση, γιατί υπάρχουν πολύ άγνωστοι χοί προς το παρόν. Δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα κονδύλια του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και του Ταμείου Εγγύσεων. Θέλουμε στην πρώτη αξιολόγηση που θα κάνουμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο ανταποκρίνεται το Ταμείο με τους στόχους, ε, στους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ώστε οι πλούσιοι να μην γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Υπάρχουν πολλά σημεία λοιπόν που δεν θα διαφύγουν τις προσοχές μας και πιο μακροπρόθεσμα μιλάω για το 2020 και μετά θα πρέπει να δούμε πού απαιτείται υψηλό κίνδυνο, γιατί είναι χρήσιμο για μερικέ δραστηριότητε, αλλά όχι για όλε. Χρειάζονται και επιδοτήσει, χρειάζονται και επιχορηγήσει και τα άλλα συστήματα στήριξη, και θα δούμε σε ποιες δραστηριότητες χρειάζεται αυτός ο επιμερισμός ε, του κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει και αργότερα. Και μετά από μια δεκαετία μπορούμε, μπορεί να καταλήξουμε σε θετική αξιολόγηση, να πήγαν όλα καλά για μερικές δραστηριότητες και άλλες να κόλλησαν κάπως στη μέση. Γιατί το χρονικό πλαίσιο είναι πολύ ευρύ το βασικό πάντως είναι τι θα διδαχθούμε από όλα αυτά, τι διδάγματα θα αντιλήσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σχεδόν πιο σημαντικό από τα δύο εργαλεία που είναι συμπληρωματικά και θα πρέπει να είναι και προσθετικά μεταξύ τους. Οπότε ελάτε μετά από ένα εξάμεινο, μετά από ένα χρόνο και μαζί με την κυρία Κρέτσου που είναι αρμόδια επιτρόπος για την περιφερειακή ανάπτυξη, να θέσουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, να δούμε πραγματικά πώ εφαρμόστηκαν όλα αυτά στην πράξη και να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα μα βήματα. Ευχαριστώ κύριε Κρέλ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ. Κύριε Μολδρέ. Οι σοσιαλιστέ πάντα υποστηρίζαν το πρόγραμμα των Ακόμα και όταν ήταν πολιτική λιτότητας. Γι' αυτό χαιρόμαστε λοιπόν που πλέον το έχουμε. Το υποστηρίζουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την αρχή. Αλλά κύριε Κατάινεν, μιλήσατε για τη χρηματοδότηση και ταχθήκατε υπέρ της πολιτικής της αγροτικής και της πολιτικής συνοχής. Ε, αυτό σας θυμά, αλλά δεν είχατε και κάποια άλλη ευκαιρία, γιατί ξέρετε ότι ο προπολογισμό της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής πολιτικής προς τα κράτη-μέλη έχει ήδη κατανεμηθεί σε ε, εθνικά μερίδια και ποτέ δεν θα είχατε συγκατάθεση και συνένεση από τα κράτη-μέλη αν το είχατε βγάλει από εκεί. Τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, μπορούν να συμφωνούν με την χρηματοδότησή σας, την πρόταση χρηματοδότησης. Δεν θα τους κοστίσει τίποτα. Γιατί δεν θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση. Η Γερμανία, τα 8 δις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αν είχε δώσει λοιπόν αυτά τα 8 δισεκατομμύρια ε, για το Επενδυτικό Ταμείο, ε, θα έχει λυθεί το μισό πρόβλημα. Δεν είναι σωστό με τον ορίζοντα 2020 να χρηματοδοτούμε τα ίδια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τον παράγοντα μειόκλευσης του Ταμείου Επενδύσεων. Στο ορίζοντα 2020 προαγάγει την ε, έρευνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και με το Connecting Europe Facility. Το ίδιο συμβαίνει. Πρόκειται για έργα τα οποία έχουμε κοιτάξει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κοιτάμε πού μπορούμε λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε έργα υποδομών. Όλα αυτά λοιπόν είναι δύσκολα και γι' αυτό λοιπόν ως Κοινοβούλιο εξακολουθούμε να προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξέρω αυτό το τριπλό α, δεν είμαι τραπεζικός, αλλά αυτό το τριπλό α όντως εξαρτάται από τα 16 δισεκατομμύρια που καλούμαστε τώρα να δώσουμε ή μήπως πρόκειται, υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Βλέπουμε δηλαδή κάποια ποσά, κοιτάμε στους αιτήσεις προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάμε τι μπορούμε να βρούμε κάθε χρόνο, γιατί τα χρήματα αυτά βρίσκονται Μπορεί να μην τα βρούμε στην αρχή, αλλά θα τα βρούμε. Δεν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε με τέτοια οδό για να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί σε ό,τι αφορά τα κονδύλια αυτά. Για τα 16 δισεκατομμύρια αυτά θα πρέπει να έλθουν κάποια στιγμή από όπου και αν προέρχονται. Αλλά θα πρέπει να επιτρέπεται να κοιτάμε σε ό,τι αφορά τέτοια δημόσια χρήματα, να δούμε τι project, τι έργα εγκρίνονται. Για να ξέρουμε ότι δεν χρηματοδοτούμε για παράδειγμα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την Ευρώπη 2020. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς ε, υπερβολική πολιτική ανάμειξη. Ίσως να κατάλαβα και λάθος αυτά που είπατε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συμμετέχει και σε ό,τι αφορά τις σημαντικές ε, εργασίες και λειτουργίες του FC. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο, από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, ποτέ δεν είναι το θεσμικό όργανο που πατάει το φρένο όταν ε, πρόκειται για επίμαχα ζητήματα, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχετε κάποια ιδέα για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται τα έργα αυτά. γιατί η Γερμανία και για άλλες χώρες υπάρχουν ε, πάρα πολύ μεγάλη κατάλογη προτινόμενων έργων, τα οποία όμως ήδη χρηματοδοτούνται. Γιατί ζητούν λοιπόν χρηματοδότηση εκ νέου. Ίσως θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κρέλα, η Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Α, συγγνώμη, από το ECR δεν βλέπω από του Δυτικού Συντονιστέ κανέναν, από του συντονιστέ, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάνκοφτσιτ από την ΑΛΤΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη Αντιπρόεδρε Κατάινεν, αξιότιμη Αντιπρόεδρε Μόλτερερ. Θα ήθελα εκ μέρους των φιλελευθέρων να σας καλωσορίσω θερμά ε, στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο και να σας ευχαριστήσω ε, για τη συνεργασία και για τη συζήτηση που είχαμε, για το χρόνο που μας αφιερώσατε κύριε Κατάινεν. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας γιατί στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική. Και η ομάδα μας η Άλντε, η Φιλελεύθερη, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την οικονομική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της απασχόλησης και μας ενδιαφέρει πολύ αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και ε, η επιτυχία αυτής της Επιτροπής, ε, της Επιτροπής Γιούγκερ και του Κοινοβουλίου θα κριθεί το 2019 με τα αποτελέσματά μας σε ό,τι αφορά το κατά πόσο καταφέραμε να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία. Από αυτή την άποψη μπορείτε να είστε βέβαιοι για την αμέριστη υποστήριξή μας. Και ελπίζω ε, η πρωτοβουλία αυτή και η μεθοδολογία που επινοήσατε να στεφθεί με επιτυχία. Εγώ είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στρατηγική στην Αδριατική και το Ιόνιο. Και υπό αυτή την ιδιότητα θα ήθελα να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Η στρατηγική ε, περιλαμβάνει την Ιταλία, τη Σλοβενία, την, ε, ε, την Ελλάδα, την Κροατία τη και υποψήφιες χώρες, Σερβία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Οχτώ είναι οι χώρες που εμπλέκονται σε αυτή την στρατηγική. Με ενδιαφέρει κυρίως ε, οι ενεργειακές, ε, με ενδιαφέρει κυρίως οι ενεργειακές υποδομές, γιατί στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδροελεκτρικής για παράδειγμα ενέργειας, και έχουμε και πολλά σχέδια για την κατασκευή σταθμών ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλβανία και στην Κροατία. Μία χώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλη δεν είναι. Έχετε σκεφτεί τη δυνατότητα αξιοποίησης της, η, της Ιταλικής αγοράς που έχει πρόβλημα με τον εφοδιασμό της ενέργειας. Δηλαδή το ΕΦΣΙ, αυτό το Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων, ε, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τέτοια προγράμματα σε χώρες μέλη και σε υποψήφιες χώρες για τις ανάγκες των χωρών μελών. Και από αυτή την άποψη ε, πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού κεφαλαίου γιατί φαντάζομαι θα είναι εν μέρη δημόσια αυτά τα προγράμματα και εν μέρη ιδιωτικά. Μπορείτε έστω και μερικώς να μου απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάκοφτσιτς, Ο κύριος... Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε Κατάινεν και κύριε Αντιπρόεδρε, μόλις ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζουμε ότι θα είναι αυτός ο διάλογος ειλικρινής και αποδοτικός. Έχω τις εξής παρατηρήσεις να σας υποβάλλω. Δεν μπορούσε κανείς συνέχεια να, να, να φιλοσοφεί τον για το Ταμείο Επενδύσεων και ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και προβάζουμε και από κάποιους συναδέλφους σε σχέση με αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα όμως βέβαια θα πρέπει τώρα πια κάτι να κάνουμε ούτως ώστε να αποδώσει αυτή η υπόθεση γιατί έχουμε εκατομμύρια ε, ανέργους που, στους οποίους το οφείλουμε, το οφείλουμε επίσης και στην Ευρώπη όλοι και στις ΜΜΕ, γιατί το πρόγραμμα Juncker βρίσκεται στην καρδιά της εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δυνατότητά της να μπορέσει να δώσει κάποιες απαντήσεις για ανάπτυξη και απασχόληση. Οπότε και έτσι θα κρυθεί η Ευρώπη αν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Οπότε έχουμε τώρα την υποχρέωση του να αναλάβουμε δράση ούτως ώστε να βγει κάτι. Είστε ενώπιον της Επιτροπής ε, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και κάπως ε, παρακολούθησα σε σχέση αυτά που συστήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή και στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών και ξέρω ακριβώς πώς βλέπετε τους στόχους της Περιφερειακής Επιτροπής και υπάρχουν εδώ πέρα κάποια ερωτηματικά τα οποία αναδύονται. Πρώτα πρώτα. Άκουσα τι είπατε, ότι δηλαδή δεν ε, υπάρχουν εδώ, δεν συντρέχουν γεωγραφικά κριτήρια. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς έχουμε διαθέσει 350 δις ούτως ώστε να εξισωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Και αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να υπάρξει συμπληρωματικότητα όσον αφορά τις ε, επενδύσεις του Ταμείου Επενδύσεων, ούτως ώστε να ε, μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους της ε, περιφερειακής πολιτικής. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάποιο είδους διαταραχή, γιατί υπάρχει αυτό το ρίσκο, μια που οι επενδυτές θέλουν οι επενδύσεις τους να κατευθύνονται προς τις μεγάλες Μητροπόλεις. Επομένω, η πολιτική το θέμα είναι πώ θα μπορέσει να δώσει ένα τέτοιο προσανατολισμό στι επενδύσει, ώστε να κατευθυνθούν προ κάποιε περιφέρειε εκεί όπου είναι η ανεργία πάρα πολύ μεγάλη. Ε, εκεί που είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προσχόληση οι επενδύσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Οπότε Εγώ προχωρώ από την Ρεωνιόν. Είναι μια νήσος, είναι περιοχή της απότατη περιφέρειας. Το δε πλάνο Γιούγκερ σήμερα κινητοποιεί τους ε, οικονομικούς παράγοντες. Οπότε δημιουργούνται και σοβαρές ελπίδες. Όμως το χειρότερο απ' όλα είναι ε, να υπάρξει απογοήτευση μετά την ελπίδα. Γιατί πρόκειται για όλε αυτέ τι απομακρυσμένε ε, περιφέρειε, όλε αυτέ που υστερούν στην ανάπτυξη, στην απότερη περιφέρεια. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιε θα είναι οι συνέπειε τι θα γίνει σε σχέση με το πλάνο Γιούγκερ. Για πέστε μας λοιπόν την γνώμη σας. Τώρα έχω ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας αναφέρω. Για να αποδώσει αυτό μας το όραμα θέλουμε να συμμετάσχουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτές οι αρχές είναι οι πιο δόκιμες, τόσο ώστε να οργανώσουν τα οικονομικά, ούτως ώστε τα ταχαίως να βοηθήσουμε προτάσεις στην Τράπεζα Επενδύσεων. Από ό,τι, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον στη Γαλλία, προς τα εκεί πάμε, γιατί συνεργάζεται το κράτος με τις περιφέρειες, τόσο ώστε να υπάρχει επεξεργασία προτάσεων. Τρίτη παρατήρηση. Και τελευταία, με ικανοποίηση άκουσα να λέτε ότι η βασική έρευνα πρόκειται να είναι ε, επιλέξιμη για το πρόγραμμα Juncker. Πρόσφατα πήγαμε στις ε, κάτω χώρες σε σχέση με, τις, ε, με την έρευνα και την εξειδίκευση και είδαμε ότι γίνονται πολλά σε αυτόν τον τομέα. Και σας τονίζω το ότι θεωρώ ότι η λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη, η γαλάζια οικονομία είναι πολύ σημαντικέ. Το πώ μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή οι θάλασσε και οι ωκεανοί για την ανάπτυξη και σήμερα και αύριο. Ε, οι Ινδίε με αυτό κάνουν. Ε, κάνουν τρομερέ επενδύσει όσον αφορά τον Ειδικό ωκεανό και τον βυθό του Ειδικού ωκεανού. Εμεί είμαστε μια παγκόσμια δύναμη κατά θάλασσα. Οπότε θα πρέπει να δούμε την μπορούμε να κάνουμε, τόσο ώστε να ωφεληθούμε, να ωφεληθεί η Ένωση στη αυτή, αλλά επίσης και όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές, ε, τα λιμάνια τη Ένωση κλπ. Δεν θα πρέπει αυτό να το παραβλέψουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους δύο αντιπροέδρους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ε, παρουσίασή τους και για την ευκαιρία που μας δίνουν να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν είναι η πρώτη, όπως αναφέρθηκε, είχαμε διάφορες ευκαιρίες και στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια και άλλωστε έχουμε ψηφίσει στην Επιτροπή μας όπως είπατε. Θα ήθελα να τονίσω εξ ονόματος της ομάδας μου ότι φυσικά είμαστε υπέρ ενός εκτενούς προγράμματος επενδύσεων επενδύσεις, τουλάχιστον στην πραγματική οικονομία. Χρειάζονται και δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσεις για να εξέλθουμε τι κρίσεις, να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη και ω πράσινη για να κάνουμε ένα βήμα πίσω από την πολιτική λιτότητα. Χαίρομαι λοιπόν που αναφερθήκατε στην πολιτική συνοχής. Αυτό που μας απασχολεί όλους και αυτό είναι η βασική ε, κριτική των πρασίνων για την διαμόρφωση αυτού του σχεδίου επενδύσεων είναι η κοινωνική και η δημοκρατική πτυχή η οποία θεωρούμε ότι δεν τονίζεται επαρκώς στο επενδυτικό πρόγραμμα. Έχω την εντύπωση από τις ε, εμπειρίες που έχουμε στην πολιτική συνοχή και από, την, ε, από τα δραστηριστικά ταμεία ότι δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που μάθαμε. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη τη κοινωνία των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, τη τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζεται αυτό επαρκώ. Το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Επίση, ένα θέμα είναι η στοχοθεσία. Οι επενδύσει δεν είναι αυτό ο σκοπό. Ούτε κάθε επένδυση είναι καλή, εφικτή ε, και βιώσιμη ή ευκταία. Το θέμα λοιπόν είναι σε ποιους τομείς θα επενδύσουμε και ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη, τον Ευρωπαίο εργαζόμενο. Και εδώ λοιπόν να ρωτιόμαστε για το εξή. Η εξασφάλιση της τοχοθεσίας, αφενός δηλαδή, η δέσμευση για τους στόχους της Ευρώπης 2020. Δεν μιλάμε μόνο για απασχόληση και βιωσιμότητα, αλλά για καταπολέμηση της ένδυας, για προστασία του περιβάλλοντος, για ισότητα, εκπαίδευση. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σημαντικά. Είναι, έχουν σημαντικό, σημαντική θέση στην ε, στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Πώς διασφαλίζονται λοιπόν αυτές οι επενδύσεις και οι κοινωνικές επενδύσεις. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν Αγαπητέ Αντιπρόεδρε Μόλτερερ, πού λοιπόν διασφαλίζεται αυτό ότι ακόμα και ένα τέτοιο σέντερ θα ταπανηθεί σε δομές ε, για την εκπαίδευση, για την αγορά εργασίας, για κοινωνικές επενδύσεις. Ξέρω για παράδειγμα από την Επιτροπή Απασχόλησης ότι υπάρχει μια πολύ έντονη συζήτηση ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι στον τομέα ε, της ε, απασχόληση στην ε, Διοικητική Επιτροπή που θα επιλέξει τα έργα προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση ότι θα λεφτούν υπόψη ε, αυτές οι πτυχέ. Αλλά δεν προβλέπονται ποσοστώσεις. Οι προσωρινοί κατάλογοι των κρατών μελών μας οδηγούν να πιστέψουμε ότι περιλαμβάνεται πάρα πολύ ελλειπώς αυτή η κοινωνική πτυχή. Πολύ λοιπόν ανησυχούμε ως πράσινοι. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα όμορφα λόγια θα μετατραπούν σε πράξεις, θα υπάρχουν ουσιαστικές επενδύσεις. Και οι επενδύσεις δεν είναι αντίθετες με την Ευρώπη 2020. Για παράδειγμα στο θέμα του κλίματος. Να μην υπάρξουν επενδύσεις σε πυρηνικά, σε οδικές μεταφορές, για τις περιφερειακές ποσοστώσεις τώρα. Ξέρετε όλες, ξέρετε όλες τις μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την δυναμικό απασχόλησης του ΕΦΣΥ που θα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο αν υπάρξουν επενδύσεις σε περιφερειές με υψηλή ανεργία. Και εφόσον γίνουν σημαντικές αλλαγές και ληφθούν σημαντικά μέτρα στα κράτη-μέλη, πώς λοιπόν διασφαλίσετε αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο, η κυρία Νταματώ. Κομισάριο Ευχαριστούμε κύριε Πίτρο που ήρθατε εδώ. Είπατε ότι χρειαζόμαστε κατηρτισμένους ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση της απασχόλησης αλλά και της ανάπτυξης θα πρέπει βέβαια να γίνουν κάποιες δαπάνες πέραν και εκτός των ε, ελλημάτων και ε, του, του χρέους όπως είπατε και εσείς. Και είπατε επίσης ότι χρειάζεται μία ανάπτυξη που όμως να καλύψει και τις κοινωνικές ανάγκες. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από τα διορθωτικά ταμεία και αυτό να λυθεί υπόψη στην υπολογισμό του ελλείμματος. Θα πρέπει κάτι να γίνει για τις ανισότητες που στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτό το ταμείο θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη. Να, ως παράδειγμα, ε, έχει σχέση με το κοινωνικό ταμείο. Ξέρουμε ότι μόνο λίγα κράτη δείχνουν ευελιξία σε σχέση με το ΕΦΣΙ. Αλλά, αλλά όμως το κοινωνικό ταμείο είναι τελείως διαφορετικό και όσον αφορά τον στόχο και όσον αφορά τη λογική τους. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πέντε ακόμα ονόματα στον κατάλογο των ομιλητών. Να θέσετε παρακαλώ πολύ σύντομες ερωτήσεις για να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις απαντήσεις ε, των ε, προσκεκλημένων. Κύριε Σπυράκη. Well, uh, I think that the question is for both. Νομίζω ότι το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο, και στον Αντιπρόεδρο Κατάινεν και στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να σας ρωτήσω κατά πόσο η Επενδυτική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση, αλλά αν θα πάρουν ε, υπόψη, πέρα από τη βιωσιμότητα του έργου, τις ειδικές ε, ε, συνθήκες που επικρατούν, οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες όπως η Ελλάδα. Και το θέμα είναι κατά πόσον το ΕΦΣΥ θα μπορέσει να αναλάβει τον κίνδυνο αυτό και να καλύψει τον κίνδυνο αυτό. Δεύτερη ερώτηση, σε κατά πόσον στην ε, διαδικασία επιλογής των έργων θα ληφθεί υπόψη η βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν με το σχέδιο Juncker. Κατά πόσον θα επικρατήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Βέσο. Κύριε Μπράσο, παρακαλώ να είστε σύντομα. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται με αυτή την πλατφόρμα των επενδύσεων για να καταλάβουμε καλύτερα, αν κατάλαβα καλά. Πρόκειται για πλατφόρμες χρηματοδότησης που μαζεύουν πόρους και κατόπιν ε, συντονίζουν ε, τις επενδύσεις. Ε, κατ' εσάς, είναι δυνατόν στο εσωτερικό αυτής της πλατφόρμας να υπάρχουν και εγγυήσεις χρηματοδότησης των projects που έχουν απότματα θετικά αλλά μπορεί βράχει πρόθεσμα να μην είναι πάρα πολύ αποδοτικά όπως πολλές φορές συμβαίνει με άλλες επενδύσεις. Επομένως ε, θα, πρέπει να δούμε το ότι μπορεί να έχουμε κάποιες ε, εξωτερικότητες όπως λέμε που μπορεί να ωφελούν άλλες ε, επενδύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι περισσότερες παρατηρήσει αφορούσαν τι θέσει τη επιτροπή προπολογισμών. Φαντάζεστε, το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή προπολογισμών. Και το πιο ζήτημα είναι από πού θα πρέπει να προέλθουν τα κονδύλια. Δεν πρόκειται να την ξαναθέσω αυτήν την ερώτηση γιατί θα ανοίξω το κούδι τη Πανδώρα. Προσπα... Προτιμώ να την αποφύγω. Ερωτώ ποια είναι η σχέση των διαρθρωτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί Βλέπουμε στα έγγραφα ότι δεν υπάρχει μηχανισμός ε, για το κατά πόσο τα ε, διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο του ΕΦΣΥ. Άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν. Αλλά υπάρχει δυνατότητα ε, συνδυασμού των επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων με τις επενδύσεις του στρατηγικού ταμείου. Μπορείτε να μας τα πείτε αυτά με απλά λόγια έχουμε το ταμείο και οι ιδιώτες επενδυτές έρχονται χωρίς πολιτική επιρροή, υποτεθήστο, χωρίς γεωγραφική επιρροή, χωρίς γεωγραφική κατανοή. Πολύ σημαντικές αυτές οι δύο επιρροές, η πολιτική και η γεωγραφική. Οπότε έρχονται οι επενδυτές από διάφορα μέρη με σχέδια υψηλού κινδύνου, θέλουν εγγύησεις, καλές εγγύησεις από το σύστημα εγγύσεων και αρχίζουν να οργανώνουν τα σχέδιά τους. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Τι γίνεται με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία. Πώς θα συνεργαστούν, πώς θα ε, συνδεθούν με το ΕΦΣΥ. Επίσης, ε, η κυρία Μπρέσο ρώτησε για τις πλατφόρμες. Είναι συναφές αυτό το ερώτημα. Γιατί έχουμε δύο εκδοχές εδώ. Η μία είναι ε, ξεχωριστά τα διαρθρωτικά ταμεία από το ΕΦΣΥ και η δεύτερη εκδοχή λέει συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΦΣΥ. Κύριος Βαρμίλτεμπορκ, πολύ σύντομα. Μία ερώτηση για τα κριτήρια επιλογής. Ε, μιλήστε για εταιρείε με 2-3 ε, εργαζόμενους, αλλά και μεγάλες εταιρείε έχουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Και ακριβώς επειδή μεγάλες επιχειρήσεις ε, ωφελούν και τις μικρότερες, γιατί λάβατε αυτή την αυθαίρετη απόφαση να βάλετε ένα όριο στους 3.000 ε, εργαζόμενους σε μία επιχείρηση, αποκλείοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, από τη δυνατότητα να υποφεληθούν από τις ε, εγγύησεις. Κύριε Μπόμποβιτς, παρακαλώ σύντομα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την ιδέα αυτή γιατί πιστεύουμε ότι η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα εξαρτηθεί από το έργο αυτό, από το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία. Οι Εθνικέ Τράπεζε Επενδύσεων, για πείτε μα, τι ρόλο θα δραματίσουν ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεύτερη ερώτηση. Υποστηρίζω αυτό που είπε ο κύριο Γιάκοπτσιτ, ότι θα πρέπει να βρούμε κοινά έργα σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Τριατική και το τροματικό σταθμό φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα επιλύσουμε περιβαλλοντικά ζητήματα στη Βόρεια Τριατική και θα κάνουμε ένα βήμα προς την Ενεργειακή Ένωση. Και τρίτον, είμαι από τη Σλοβενία εγώ. Είχαμε πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την προστασία από πλημμύρες θα μπορούσε το ΕΦΣΙ να χρησιμοποιηθεί επιπροσθέτως προς το ταμείο το οποίο χρησιμοποιούμε για την προστασία κατά των πλημμυρών. Τα πιο πολλά κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Συνοχής. Θα μπορούσε να συμπληρώσει το ΕΦΣΙ. Δεν υπάρχει οικονομική απόδοση στην περίπτωση αυτή. Αλλά γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ότι η δράση εκ των υστέρων σε περίπτωση πλημμύρα που δημιουργεί ζημιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Δυστυχώ θα πρέπει να. Δεν μπορούμε να ακούσουμε άλλε ερωτήσει για να δώσουμε ευκαιρία στου προσκεκλημένου μα να απαντήσουν. Ελπίζω να μην είναι η τελευταία άλλωστε συζήτηση που θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε. Έχουμε εκφράσει ήδη την επιθυμία μα αυτή και ελπίζουμε να βλεπόμαστε σε τακτικά διαστήματα προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Ο κ. Κατάνη να ξεκινήσει. Πρέπει να σας τα πω πάρα πολύ σύντομα γιατί έχω μια άλλη υποχρέωση στη συνέχεια. Πρώτα πρώτα το μήκος των επενδύσεων δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Επομένως είναι λογικό κανείς να κοιτάει το τι θα γίνει. Γιατί έχουμε 60 δις σε τρία χρόνια. Ε, από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χτες διάθεσε 75 δις ετησίως. Έχουμε 8 σχολεία στο Μέλλον Βασίλειο, Οπότε πάρα πολλέ από αυτές τις ανάγκες που αναφέρθηκαν εδώ ταιριάζουν στην καθημερινή δουλειά, ρουτίνα τη Τράπεζα επενδύσεων. Γιατί τώρα μιλάμε όμως για ένα εργαλείο πολύ διαφορετικό. Πρώτα-πρώτα, ότι άλλε επιλογέ υπάρχουν. Αν δείτε τι γίνεται με το κεφάλαιο 1α, έχουμε το, το, το, το ρίζο να καλύπτει κατά 70% μόνο ο Γαλιλαίος και ο έρασμο είναι απ' έξω. Από αν αρχίσουμε τι διαπραγματεύσει με 28 κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τα τα ταμεία ή την αγροτική πολιτική, τι θα γίνει. Δύσκολα θα γίνει το πράγματα. Για την επιστολική αξιολόγηση η Standard Poor's ήδη μας έχει υποβαθμίσει. Και είναι αλήθεια έχουμε 25 εκατομμύρια ε, ο, οφειλές. Και δεν θυμάμαι πόσο άλλο, πόσο άλλο υπάρχουν από άλλα κεφάλαια του προπολισμού. Οπότε έτσι κινδυνεύουμε να μην έχουμε τα 60 δις γιατί αυτό θα ήταν επιχείρημα να υποθυμιστεί παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάποια άλλη εταιρεία αξιολόγησης. Θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα σε κάποιες χώρες που έχουν στριμωχθεί, οπότε πολύ σοβαρό και γι' αυτό είπα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το από πού προέρχονται τα χρήματα. Βασική έρευνα και χρηματοοικονομικά εργαλεία στο ορίζον 2020 έχουμε 77 δις. Δηλαδή 48% περισσότερο από πριν από δύο χρόνια είχαμε. Είπαμε ότι τώρα με αυτά τα οικονομικά εργαλεία θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα. Όπως σας είπα, έχω πάει σε μια σειρά πανεπιστημίων που, που τα χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία και που προτίθενται τώρα να τα, χρησιμοποιήσουν τα, ε, και στο μέλλον, ακόμα και στην Κύπρο που είναι και αυτή η χώρα στριμωγμένη οικονομικά και γνωρίζουν ότι θέλει ο ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει, αλλά και οι κυβερνήσει. Δεν μπορούν όμω να προσπαθούν δάνεια. Στην Κύπρο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επομένω, α κρατήσουμε μια ανοιχτή στάση, γιατί έτσι θα βοηθηθεί η έρευνα αν έχουμε τα χρήματα. Κύριε Μαρζέ, αναφέρατε ότι οι πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τους τομείς όπου υπάρχει πρόβλημα απασχόλησης. Ναι, θα γίνει και αυτό. Αλλά ας πούμε να κοιτάξετε τι γίνεται στις ΜΜΕ. Πάντοτε το ίδιο είναι το πρόβλημα. Στη Γαλλία, στην Γερμανία, στην Κύπρο, παντού. Εκεί δεν υπάρχει το κεφάλαιο, δεν υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεν είναι θέμα γεωγραφικό. Επίσης έρευνα, υποδομές. Γίνεται αυτό στα πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε όμως επενδύσεις σε κάποιες στοχότερες περιοχές για να μπορέσουμε να δώσουμε μια στροφή προς την ανάπτυξη. Και παρά δεν υπάρχει προδιάθεση χρημάτων στο ΕΦΣΙ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στο ότι θα πρέπει διαφορετικά εργαλεία να χρησιμοποιηθούν σε άλλο μέρος στην Ευρώπη για, για το, σκοπό που θέλουμε σε κάθε μέρος. Γι' αυτό και είπαμε ότι αυτός ο κόμβος συμβουλών είναι πολύ σημαντικός, ρόλο και όλες οι χώρες να μπορέσουν να ωφεληθούν. Υπάρχει επομένω η τεχνική ε, αρρωγή ευρωπαϊκής κομισιών που θα βοηθήσει και τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, περιοχές και έτσι να ωφεληθούν από το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Κυρία Ντεμάτο. Έγινε κάποια παρεξήγηση μάλλον. Δεν είπα να κόψουμε τα χρήματα της παιδείας ε, λόγω του ελλείμματος. Το χρηστούν κανόνα. Ναι, ε, βέβαια και αυτές όλες οι δαπάνες να μην μετρήσουν για έρευνα και παιδεία. Αλλά τότε θα πρέπει να βγάλουμε και να μην συνυπολογίσουμε και όλα τα κονδύλια του προπολογισμού. Και γι' αυτό είπα ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κρατικό χρήμα για να εθαρρύνουμε τα κρατημέλη να δαπανίσουν περισσότερα ή να φουσκώσει έτσι το χρέος. Και αυτό και είπαμε να θέλουμε να ελκύσουμε πόρους και να προέλθουν αυτοί οι πόροι στο εγγυσμένων από τον ιδιωτικό τομέα. Κυρία Σπυράκη, το ΕΦΣΙ καλύπτει αυτούς τους κινδύνους. Τις πρώτες συνέντησα κάποιους ε, εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και εξηγήσαμε ότι θα καλυφθεί ο κίνδυνος από το ΕΦΣΙ όπου υπάρχει ο κίνδυνος. Σε άλλες χώρες θα καλύψει και άλλους. Εδώ θα... Σας ευχαριστώ. Κύριε Μόλτερερ, εν συντομία. Κύριε Βανίλστερόι, έχουμε εμπειρία με δανειοδότηση κεντρικών κονδυλίων ε, τα project bonds, τα ομόλογα έργου. Το κάνουμε. Αλλά έχουμε και αποκεντρωμένα κονδύλια ε, βλέπε πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πρωτοστατεί εδώ η Ισπανία. Η Μάλτα και η Πορτογαλία επίσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτό το μηχανισμό. Και για να σας δώσω μια γεύση, από το 2007 μέχρι το 2013 90 ε, δισεκατομμύρια τα δώσαμε για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών ταμείων. Ήδη κάνουμε πολλά δηλαδή για τη συνοχή. Δεύτερον, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν αντικαθιστά, δεν υποκαθιστά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και το ΕΦΣΙ θα μας δώσει επιπλέον δυνατότητες για δράση. Κυρία Κρέλ, το βασικό θέμα των εγγύσεων είναι το εξής. Αν ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, αναλαμβάνουμε την ευθύνη στα λογιστικά μας βιβλία για όλη τη διάρκεια της επένδυσης που για υποδομές μπορεί να είναι δεκαετή η διάρκεια 20 ετής έως και 30 ετής. Οπότε χρειαζόμαστε τη βεβαιότητα ότι αν ξεκινήσουμε το εγχείρημα η εγγύηση θα είναι πλήρως διαθέσιμη. Αν δημιουργήσουμε την εντύπωση στον έξω κόσμο και στους ιδιώτες επενδυτές αλλά και στους οίκους αξιολόγησης ότι το θέμα της εγκυρότητας ε, της εγγύης θα κρυθεί από αποφάσεις που θα, κάθε χρόνο, θα λαμβάνονται κάθε χρόνο δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Γι' αυτό εμένουμε πεισματικά σε αυτή την αρχή και σας ζητούμε να μας στηρίξετε. Γιατί αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δεύτερον, οι πολιτικές ευρωπαϊκές Ένωσες, ε, της Πολιτικής Ένωσης είναι οι κατευθυντήριες γραμμές και για την ε, ΕΤΕΠ. Δεν βγάζουμε το κεφάλι μας. Ξέρουμε τι σημαίνει η πολιτική, στρατηγική 2020, την παρακολουθούμε. Αν δείτε τις τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ, βλέπετε ότι πριν από δεκαετίες δεν ήταν στο επίκεντρο της προσοχής ούτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε οι κλιματικές αλλαγές. Στο μεταξύ, η αποδοτικότητα των πόρων είναι το 1 τέταρτο των ε, δραστηριοτήτων μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πάνω από 1 τέταρτο των δραστηριοτήτων μας. Επιλογή των σχεδίων. Κανονική διαδικασία επιλογής που εφαρμόζει η ΕΤΕΠ και επιπλέον η Επιτροπή Επενδύσεων θα αποφασίσει να εγκρίνει ή όχι την εγγύηση για συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή η επιλογή γίνεται από επαγγελματίες και επιπλέον η Επιτροπή Επενδύσεων κρίνει κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ή όχι η εγγύηση για συγκεκριμένο σχέδιο. Κύριε Γιάκοφτσιτς, ε, Έχουμε το επενδυτικό σχέδιο ε, για τις 28 χώρε μέλη, αλλά η ΕΤΕΠ καλύπτει και δραστηριότητες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι δυνατόν να χρηματοδοτούν και διασυνοριακά ε, σχέδια. Έχουμε το μηχανισμό για τα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα. Έχουμε μηχανισμούς, facilities, διευκολύνσεις που έχουν και διασυνοριακή διάσταση. Αλλά αρχικά το ΕΦΣΙ έχει σχεδιαστεί μόνο για τι 28 χώρε μέλη. Το θέμα πολιτικής συνοχής και Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Το αντίθετο ισχύει. Είναι ένα επιπλέον όργανο αυτό, ένα επιπλέον εργαλείο. Δύο παραδείγματα. Για τι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας δεν χρειάζεται τίποτα αν συνδυάσετε δύο μεγάλες πόλεις. Γιατί οι επενδύσει αυτές θα γίνουν από του ιδιώτες, οπότε δημιουργείται το εισόδημα. Αν όμω μιλάμε για ευρυζωνικότητα στην Ήπεθρο, στι αγροτικέ ζώνε, τότε χρειάζεται ειδικό μέσο στήριξη για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Άρχισα τι συζητήσει με τον Φιλ Χόγκαν, τον αρμόδιο επίτροπο Γεωργία, για το θέμα τη ανάπτυξη τη Ήπεθρου, που είναι σημαντικό δυνητικό εργαλείο και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Και επίση με την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ ε, γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία θα ενισχύσει το δυναμικό μας. Εθνικά, εθνικοί θεσμοί πρόθεσης. Εσκεμένα χρησιμοποίησα το ρόλο, το, τον όρο θεσμοί πρόθεσης, γιατί δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη εθνικές τράπεζες πρόθεσης. Οπότε άμα πούμε εθνικές τράπεζες πρόθεσης θα αποκλείσουμε κράτη-μέλη που δεν έχουν τράπεζες, αλλά θεσμούς πρόθεσης. Πάντως ήδη χρησιμοποιούμε ε, αυτούς τους θεσμούς ε, ως μεσάζοντες για να δανείσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εθνικές συνεισφορές ε, σε σχέδια ή σε επενδυτικές πλατφόρμες. Πολύ ενδιαφέρον και δυνητικός εταίρος συνεργασίας αυτές, αυτή η θεσμή πρόθεσης. Επίσης, η ΕΤΕΠ δεν, δεν φτιάχνει, δεν κατασκευάζει σχέδια. Τα χρηματοδοτεί. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν ε, επαγγελματίες ε, επιτόπου για τη διαχείριση για την υποβολή και διαχείριση αυτών των σχεδίων. Επίσης μας ενδιαφέρει και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να αντιληφθούν και αυτές το δυναμικό συνεργασίας με την ΕΤΕΠ. Αυτό που είπε ο Ζανκλώτ Γιονκέρ όταν ε, εγγενίασε πέρυσι την πρωτοβουλία είναι ότι το ΕΦΣΙ είναι ένα τμήμα της στρατηγικής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ένα τμήμα της στρατηγικής. Η ενιαία αγορά ενεργειακής ένωσης, ε, ενέργειας ή η, η, η ενιαία αγορά κεφαλαίων είναι άλλα στοιχεία. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις το ίδιο. Αλλά με ενημέρωση, με συζητήσει μπορούμε να σας πείσουμε, πιστεύω. Και καλό θα ήταν τακτικά να έχουμε τέτοιες ανταλλαγές απόψεων, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία. Και το παράδειγμα των υποδομών που σας ανέφερα δείχνει ότι η δραστηριότητά μας επεκτείνεται εξαπλώνεται όλο και περισσότερο από ό,τι αρχικά φανταζόσασταν ακόμη κι εσείς. υποδομές είναι ένα παράδειγμα, η καινοτομία άλλο παράδειγμα. Το θέμα της ε, πληροφορίας επίσης το ίδιο. Ήδη χρηματοδοτούμε ε, εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμε πανεπιστήμια. Αυτά, μπορούμε, αυτά τα κάνουμε ήδη και με το ΕΦΣΥ μπορούμε να τα κάνουμε ακόμη και περισσότερα. Τώρα, συνεργασία του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και των Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων. Ε, μία δυνατότητα συνεργασία είναι οι επενδυτικέ πλατφόρμες. Η πρωτοβουλία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δίνει άλλη δυνατότητα συνεργασία. Και με το Compass, με τι άλλε γενικέ διευθύνσει, διανοίγεται και ένα τρίτο επίπεδο συνεργασία. Επίση, ε, δεν έχουμε αποκλείσει τι μεγάλε επιχείρησει. Ήδη χρηματοδοτούμε και μεγάλε επιχειρήσει. Απλώ λέμε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων επικεντρώνεται στι μικρομεσαίε και στι μεσαίε κεφαλαιοποίησει επιχειρήσει. Αλλά έχουμε και θέμα, προγράμματα έρευνα και ανάπτυξη για τι μεγάλε εταιρείε αλλά κυρίως οι μικρομεσαίες και οι μεσαίες κεφαλαιοποίησεις εταιρείε χρήζουν στήριξη. Γιατί οι μεγάλες εταιρείε έχουν ρευστότητα, έχουν εμπειρία, έχουν πρόσβαση στις κεφαλαγορές, κάτι που στερούνται οι μικρομεσαίες και μεσαίες κεφαλαιοποιήσει επιχειρήσεις. Τώρα, αντιπλημμυρική προστασία, την κάνουμε σε πολλές χώρες. Εκεί συνδυάζουμε τα διαφορετικά ταμεία με τα δικά μας δάνεια, τα δάνεια της ΕΤΕΠ. Μία όμως ε, σαφής προϋπόθεση, και αυτή είναι η εμπειρία μου από την προηγούμενη μου σταδιοδρομία, για την αντιπλημμυρική προστασία χρειάζεται στρατηγική στη χώρα. Αλλιώς ε, γίνεται κατάχρηση των κονδύλων. Δηλαδή επενδύουμε σε ένα τομέα και χάνουμε σε άλλο τομέα. Δημιουργούνται αντιφάσεις. Και εδώ είμαστε σκληροί και αμήλικτοι. Θέλουμε φυσικά να στηρίξουμε, αλλά ο ρόλος μας μερικές φορές είναι να πούμε και όχι για να αποφευθεί κακή διαχείριση, ε, κακή επένδυση ή κακή χρήση πόρων. Ε, γιατί είμαστε τράπεζα, θέλουμε ε, απόδοση και επιστροφή των κονδυλίων μας και γι' αυτό υγιή από επενδυτική λογική σχέδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των μελών της Επιτροπής μας και θα σας προσκαλέσουμε πάλι σύντομα. Ένα λεπτό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Παρακαλώ, ησυχία. Και συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση πρωτοβουλίας για την πολιτική συνοχή και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Η συγγήτριά μας, η κυρία Ρέινκε, η οποία κατέθεσε το σχέδιο έκθεση. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο για να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή των απόψεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε ακόμα σχέδιο έκθεσης, έχουμε ένα έγγραφο εργασία στη δημιουργούσα το οποίο κατανεμήθηκε, διανεμήθηκε. Να μιλήσω λίγο για το πώς προέκυψε αυτή η έκθεση. Ξέρετε ότι τη νέα περίοδο 2014-2020 οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις προτεραιοποιημένες κοινότητες σε όλα τα επίπεδα ως ομάδα στόχο. Με την έκθεση λοιπόν αυτή θέλουμε ακριβώς αυτό να κάνουμε, να δούμε στη φάση εφαρμογής της αρχής αυτής τι συνέβη. Αναφέρθηκαμε λοιπόν στις προτεραιοποιημένες ομάδες, ήδη από το 2009 γίνεται σχετική αναφορά. τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τώρα λοιπόν θέλουμε να δίνουμε αν υπάρχει όντως προστιθέμενη αξία. Σε καιρούς κρίσης βλέπουμε ε, ότι οι περιθωριοποιημένες κοινότητες πλήττονται ακόμα πιο πολύ από ότι οι υπόλοιπε και ιδιαίτερα ο πληθυσμό στις ε, κοινότητες αυτές ε, υποφέρει ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική για να απαλληλθούν αυτές οι συνέπειες. Εκ παραλλήλου, πολλοί δήμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα και αυτό δεν τους επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις να διοργανώσουν συνολικές πολιτικές για θέματα συνοχής σε δημοτικό επίπεδο. Η έκθεση λοιπόν θέλει να καταγράψει όλες αυτές τις καταστάσεις, να δούμε τις συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υπάρξει μια πολιτική συνοχή που θα ωφελεί πραγματικά τι προεθρεπημένε κοινότητε. Τι κάνουμε λοιπόν στο έγγραφο εργασία, το οποίο έχετε μπροστά σα. Κοιτάξαμε τι συμφωνίε εταιρική σχέση και τα λειτουργικά προγράμματα τα οποία ήδη έχουν εφαρμοστεί. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίε από το επίπεδο εργασίας όλων των θεσμικών οργάνων και προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε και την κοινωνία των πολιτών όσο πιο πολλές ομάδες γινόταν που εργάζονται για θέματα, πάνω σε θέματα πολιτικής συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ζήτημα για μας και μιλήσαμε και με εκπροσώπους περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να προσθέσουμε και την πόλη από την οποία προέρχομαι, Γέννησεν Κυρίχεν και μερικοί άλλοι δήμοι κοντινοί που συμπεριλήφθησαν γιατί αντιμετωπίζουν μεγάλη ροή μετανάστευσης ε, με μεγάλη, μεγάλα ποσοστά πληθυσμού Ρωμά για παράδειγμα που αποτελούν περιθωριοποιημένες κοινότητες. Για θέματα περιεχομένου τώρα. Μιλάμε για περιθωριοποιημένες κοινότητες, περιθωριοποιημένες ομάδες στην αρχή της συζήτησής μας συζητούσαμε έντονα το κατά πόσο θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σαφής ορισμός, το τι εννοείται με τον όρο αυτό. Τελικά επιλέξαμε την εξή λύση. Δεν θέλουμε να έχουμε πολύ στενό ορισμό του τι εννοείται. Προτιμάμε να ορίσουμε κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, υγεία, ε, βιωτικό επίπεδο. Και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν αυτέ οι ομάδε. Για παράδειγμα, το γεγονό ότι αποκλείονται από κάποιε συγκεκριμένε δραστηριότητε τη κοινωνία. Οι γενικέ αρχέ που θέλουμε να εφαρμόσουμε σε όλη την έκθεση είναι η μη διακρατική μεταχείριση και ο απότερο στόχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη ε, κατάργηση συστηματικών αιτιών ανισοτήτων. Οι ανισότητε είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Μία από τις ομάδες που συζητιέται έντονα είναι η Ρωμά στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Άρα στην έκθεση θέλουμε να κοιτάξουμε την οτροπία του ρατσισμού εις βάρος τσιγκάνων σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε γενικώ όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά αυτές τις διεκτικές μεταχειρήσεις ε, της αφιγκονοφοβίας. Ύστερα, πρόσβαση σε κοινοφιλείς υπηρεσίες από πλευρά των πληθυροποιημένων κοινωνιτήτων. Θέλουμε να μην κοιτάμε μόνο την πλευρά της ζήτησης, αλλά να κοιτάμε και αυτό που ονομάζουμε μια υπηρεσία που υποδέχεται εγκάρδια τον πολίτη. Γιατί οι κοινότητες αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε τέτοιε υπηρεσίες. Άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, όπω ανέφερα και προηγουμένω στις εργασίε μας, αλλά και για την ε, συμπερίληψη των περιφερειών επιμενοκοινωτήτων στην πολιτική συνεχή, είναι η αρχή της εταιρική σχέσης ε, με, ε, σε υποχρεωτική βάση. Η πρόσβαση στι κρυφολείς υπηρεσίες, όπως σα είπα, αποτελεί μια προσέγγιση που είναι ρετή αλλά όχι αποκλειστική στοχοθετημένες ενέργειες που ωφελούν τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, αλλά σε τελική ανάλυση ωφελούν όλη την κοινωνία, ανισχύοντας για παράδειγμα τις ε, δημόσιες υπηρεσίες. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στην έκθεση είναι η καταπολέμηση <coughs> της διαφθοράς και της απάτης στη χρήση των πόρων. Όταν ε, σε κάποιες περιπτώσεις υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται κονδύλια ε, για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αυτό έχει αποτελέσει πρόβλημα στο παρελθόν και θα θέλαμε να κάνουμε συστάσεις για τη βελτίωση αυτού του φαινομένου. Η δομή της έκθεσης θα ακολουθεί την δομή των διαφόρων φάσεων της πολιτικής συνοχής. Την προετοιμασία της ε, πολιτικής συνοχής θέλουμε να δούμε πώς γίνεται η διαπραγμάτευση των συμβάσεων εταιρική σχέση. Στη φάση αυτή για την προγραμματική περίοδο την ε, τρέχουσα έχει περάσει αυτή η φάση. Κοιτώντα λοιπόν τι ε, συμβάσει εταιρικών σχέσεων, ε, εταιρικής σχέσης, βλέπουμε ότι δεν έχει καν εφαρμοστεί αυτό από κάποια, κάποια από κράτη-μέλη για περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στην επόμενη περίοδο. Κάτι άλλο. Η αρχή ιατρικής σχέσης εφαρμόζεται σε όλη τη φάση της προετοιμασίας και ο κώδικας δεοντολογίας δεν είναι καν γνωστό ε, στις κυβερνήσεις ε, και στις αρχές σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό το διαπιστώσαμε από συζητήσεις με ΜΚΟ. Αυτό ασφαλώς αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει να το τονίσουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κατά την προετοιμασία της κατανομής των πόρων του Ταμείου συνοχή εφαρμόζονται οι αρχιετερικοί σχέσεις και ότι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ιδιαιτέρω δε από τις περιφερειμένες κοινότητε. στη φάση της εφαρμογής. Από τις συζητήσει που κάναμε προέκυψε ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση. Έχουμε δει πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα, όπου λήφθησαν υπόψη διάφορες πτυχές, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα κονδύλια από διαφορετικά ταμεία μαζί, για να υπάρξουν έργα με την ε, ενοποιημένη αυτή προσέγγιση και απασχόληση, παιδεία, στέγαση και υγεία. Είναι τέσσερις τομείς οι οποίοι συζητήθηκαν πιο πολύ. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν διάφορα ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα θέλαμε να συστήσουμε κάποια εργαλεία με τα οποία είχαμε πολύ θετικέ εμπειρίες, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη με, μέσω της κοινότητας, για παράδειγμα, που έχουν δείξει αποτελέσματα για τις περιτροπημένες κοινότητες. Κάτι άλλο που θέλαμε να τονίσουμε στην έκθεση, το θέμα της ανάπτυξης δυναμικού και ικανοτήτων. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει αμέλεια για τη συμπερίληψη ε, των κοινοτήτων αυτών, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, αλλά αυτό σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται και σε έλλειψη προσωπικού από πλευράς των αρχών. Θέλουμε λοιπόν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο να υπάρξει βελτίωση. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε ιδιαίτερω για το έγγραφο εργασία είναι το θέμα του mainstreaming. Του να ενταχθεί αυτό δηλαδή σε όλους τους τομείς. Να μην είναι μόνο στο άρθρο 9,2 των διατάξεων, αλλά να παίξει ρόλο σε, και στις υπόλοιπες διατάξει της πολιτικής συνοχής. Θεωρούμε ότι είναι οριζόντιο και εγκάρσιο το θέμα αυτό. και μπορεί να ωφελήσει όλους τους τομείς της ε, πολιτικής συνοχής. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει έλλειψη επιτυχών έργων είναι τα έργα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Πολλά project που εφαρμόζονται σήμερα δεν είναι βιώσιμα. Μετά από χρηματοδότηση δύο-τριών ετών τα project δεν επιζούν τελικά δεν επιβιώνουν. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικές συνοχής αυτής. Η περίοδος παρακολούθησης επίσης έχει φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί βλέπουμε ότι στη σημερινή φάση, στη σημερινή... σήμερα τα... η παρακολούθηση αυτή δεν γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο. Ουσιαστικά τσεκάρουμε κάποια παιδεία. Είναι μόνο προσωπική στη φύση της. Δεν υπάρχει ο ποιοτικός παράγοντας. Δεν ε, κοιτάμε κατά πόσον υπάρχει βιωσιμότητα στα έργα. Άρα πολλά μπορούν να γίνουν στον τομέα της παρακολούθησης. Και επίσης στην παρακολούθηση, θεωρούμε ότι θα πρέπει στις σχετικές επιτροπές να συμμετέχουν και οι περιφερειοποιημένες κοινότητες. Γιατί μόνο οι εκπρόσωποι των κοινότητων αυτών μπορούν πραγματικά να αποφανθούν για το πώς επηρέασε το έργο το εκάστοτε της κοινότητες τους. Τελευταίο θέμα το οποίο ήθελα να τονίσω στην έκθεση, η ανάγκη δικτύωσης. Στην παρούσα φάση βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη Εμπειρία. Και πραγματικά θα χρειαζόταν ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να μπορέσουν οι κοινότητες αυτές να μπορούν να έχουν πιο έντονο ρόλο στην πολιτική συνοχή. Όπως βλέπετε, μας ε, απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Έχουμε δαπανίσει και ενέργεια και πολύ εργασία στον θέμα αυτό. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους κιότες και με τις άλλες ομάδες, με τις ΜΚΙΟ. Έχουμε πολύ τεχνογνωσία στη λέξη και θα χαρώ να λάβω σχόλια από πλευρά σας ε, προσθήκες, κριτικές. Την άλλη τρίτη θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση των Σκιώδων και προσβλέπω στις συζητήσεις μας. Σα ευχαριστώ. Έκανα λάθο είπα ότι δώσατε το σχέδιο τη έκθεση. Ήταν απλώ ένα έγγραφο εργασίας, αλλά μα είπατε τόσο διεξοδικά που νομίζω ότι είστε έτοιμοι και για την έκθεση. Να δώσω τώρα το λόγο στους και ηγητέ. Η κυρία Κόρτ, πρώτη. Ευχαριστώ. πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η ιδεολογική προσέγγιση της μελέτης και του εγγράφου εργασίας. Ε, αξιέπαινη πρωτοβουλία. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το μέχρι τώρα έργο της. Συμφωνώ με την κυρία Ρέντκε ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική προσέγγιση ε, της πολιτικής συνοχής για τέτοιου θέματα. Επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε τις επιπτώσεις ε, που έχουν κοινωτικά προγράμματα σε κοινότητες. Και θα πρέπει να ε, εντάξουμε τις περιφερειοποιημένες κοινότητες ε, γιατί στο παρελθόν δεν ήμασταν αρκετά θερμοί και ανοιχτοί απέναντι στις κοινότητες αυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χορήγηση των κονδυλίων και τη δρομολόγηση των σχεδίων. Σχεδίων που θα ανταποκρινόταν στι πραγματικέ του ανάγκε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανταπόκριση από αυτέ. Θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο άνοιγμα λοιπόν και ζέση προ κοινότητε. Επίση, μιλήστε για τι ψευδο μη οργανώσει. Το αναφέρετε στο έγγραφο. Και Είχα και εγώ τέτοια εμπειρία. Υπάρχουν τέτοιε πλαστέ μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, εικονικέ. Εμεί πρέπει να συνεργαστούμε με πραγματικέ, ε, γνήσει, ε, υπαρκτέ οργανώσεις που θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Επίσης πρέπει να συνεργαστούμε με τοπικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών και για το σχεδιασμό και για την παρακολούθηση των κοινωτικών προγραμμάτων για να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα και να δημιουργήσουμε ικανότητες η αηφορία, η βιωσιμότητα είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις και νομίζω ότι είναι και λόγος ε, ύπαρξη αυτού του προγράμματος ε, ε, εξασφάλιση της βιωσιμότητας τέτοιων σχεδίων στις περιθωριοποιημένες κοινότητες. Θα ήθελα και κάποιες διευκρινήσεις. Μερικές ήδη αρχίσετε να τις δίνετε. Αναφέρατε στο έγγραφο ότι αντί να δώσουμε ορισμό των περιθωριακών κοινοτήτων, η έκθεση θα ξεκινήσει από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πρόσβαση σε παιδεία και υγεία, ε, αλλά πιστεύω ότι έτσι θα χάσουμε μία ευκαιρία. Γιατί όταν δίνετε παραδείγματα στην, στο έγγραφό σας, μιλάτε κυρίως για τους Ρωμά. Πείτε μου λοιπόν, πόσο μπορούμε να διευρύνουμε τα παραδείγματα Επίσης η έκθεση είναι ευκαιρία να στραφούμε σε πολιτιστικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και θα περιορίσουν τον αποκλεισμό ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Επίσης ε, προσοχή στους ε, ευάλωτους νέους, ε, στους αναπήρους, στα παιδιά ή σε όσους είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της φτώχειας. Να μην ξεχνάμε επίσης και τις περιφερειακές και αγροτικές κοινότητες. Αυτά και προσβλέπω σε στενή συνεργασία με την εισηγήτρια. Πάρα πολύ. Αν τώρα και οι υπόλοιποι σκέψεις το λόγο, βλέπω να ζητάει ο κύριος Γιάκοβτσιτς. Ευχαριστώ. Μόλις πριν από λίγο είδα το έγγραφο. Το φιλομέτρησα γρήγορα και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το, το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα της κοινότητας Ρωμά στην Ευρώπη. Και μάλιστα ε, το ανέφερα και στην Ολομέλεια. Είμαι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα προβλήματα της κοινότητας των Ρωμά. Γιατί ως πρόεδρος της ε, Ίστριας, της επαρχίας της Ίστρας για 20 χρόνια. Είχα μεγάλη συνεργασία ε, με την κοινότητα των Ρωμά και γνωρίζω τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης που αντιμετωπίζουν. Καλογραμμένο το έγγραφο και σίγουρα είναι σημαντικό αυτό το θέμα και γι' αυτό αποφάσισε να το θέσει στο επίκεντρο της έκθεσης της η συνάδελφος από τους Πρασίνους. Βέβαια, δυστυχώς η Ρωμά δεν είναι η μόνη περιθωριοποιημένη κοινότητα στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο, να, να περιλάβουμε και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες. Οι, οι άποροι, για παράδειγμα, οι άστεγοι Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πρόσφατα με εκπροσώπους ε, της Ένωσης Αστέγων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή πρόβλημα με τους Αφρικανούς ε, μετανάστες. Ε, πρόβλημα αντιμετωπίζουν κυρίως οι μεσογειακές χώρες, αλλά έχουμε και άλλες κοινότητες περιθωριοποιημένες, οπότε η συζήτηση δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στους Ρωμά γιατί το 95% του εγγράφου αφιερώνεται στους Ρωμά. Σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτή την κοινότητα, αλλά έχουμε ήδη πολλές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν τους Ρωμά και στηρίζουν τους Ρωμά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η έκθεσή μας είναι έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μην δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει να επεκτείνουμε κάπως το θέμα. Λυπάμαι, αλλά στην επόμενη συνεδρία δεν θα είμαι παρόν. Θα βρίσκομαι στην Κροατία, αλλά σίγουρα θα σας στείλουμε τις παρατηρήσεις μας και γραπτός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστερ αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώχιμ Ζέλερ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δεν ε, έχει την δυνατότητα να παρευρεθεί εδώ σήμερα για να μιλήσει για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το αντικαθιστώ, γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Καταφέρατε με μεγάλο ενθουσιασμό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ε, εκφραστείτε για το θέμα αυτό. Είχαμε τότε ήδη προσαρμόσει τους κανονισμούς και δώσαμε στα κάθε μέρη τη δυνατότητα να κάνουν, ε, να τα εφαρμόσουν αυτά για τις περιοχές σύγκλησης. Τώρα θέλουμε ενοποιημένη προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και αυτό να χρηματοδοτηθεί από τα ταμεία μας. Είχαμε πει τότε ότι μέχρι 6% των ταμείων, των περιφερειακών ταμείων, ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης μπορεί να ταπανηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και εκ των υστέρων ε, αποδείχθησε, αποδείχθησε ότι χρειαζόταν ε, σχέδια δράση σαν κράτο μέλο. Και αυτά που είχαμε από άποψη εργαλείων και χρηματοδότηση θα έπρεπε να ενταχθούν σε μια ενοποιημένη προσέγγιση. Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα, ποιοι ήταν τότε, ποιοι ήταν τότε οι διαφορές που προέκυψαν. Είτε μιλάμε για τους Ρωμά όχι και καλά κάνετε και μιλήσατε γιατί είναι μια αρκετή, αρκετά σημαντική ομάδα και έχουμε και στην Ολλανδία αιτήματα από οργανώσεις ε, και μιλάμε για την τοποθεσία συγκεκριμένων έργων στέγασης, για παράδειγμα, εκπαίδευσης. Και πώς γίνεται να μην ενισχύεται ο περιεθρεμένος χαρακτήρας των ομάδων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί αυτά που έχουμε πετύχει είναι μηδαμινά. Και γιατί λοιπόν γίνεται αυτό. Ούτε με το Ταμείο Συνοχή, ούτε με το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη δεν καταφέραμε να πετύχουμε αποτελέσματα επειδή δεν υπάρχει απορρόφηση, επειδή δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση από τα κράτη-μέλη. Ας το εξετάσουμε αυτό. Για να μην βρεθούμε στο ίδιο σημείο σε κάποια χρόνια. Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν στα εθνικά κράτη-μέλη και εσείς μιλάτε για territorial proximity, για περιφερειακή εγκύτητα. Πολύ καλή λύση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει καλή παρακολούθηση, καλή, καλύτερη αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης. Εμεί αυτή την αρμοδιότητα έχουμε, οι άλλε αρμοδιότητε οι άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ίσω εξετάσουν από άλλη οπτική γωνία. Μήπω θα πρέπει να τα βάλουμε κάποια πρωινή ώρα, να γίνει κάποια μεγάλη συζήτηση. Για να μην υπάρχει ανεπιθύμητο, τελικά, ανεπιθύμητη έκφραση των συζητήσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ συνάδελφε για το έργο σας. Ξεκινώ από το τέλος για να σας πω τη σκέψη μου. χρειάζεται να εμπλακούν όλοι τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές αρχές, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η υπόθεση, γιατί μιλούμε για το ότι χρειάζεται να υπάρχει προγραμματισμός και υλοποίηση αυτών των δράσεων ε, όσον αφορά τις ανάγκες των περιφερειμένων αυτών, τις οικονομικές, κοινωνικές κλπ. Και ακριβώ όπω λέτε, έχουμε αυτέ τι πρωτοβουλίε. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια χρηματοδότηση. Είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία το 2010 να συντονιστούμε όπως έγινε με το Erasmus και να χρησιμοποιήσουμε τώρα αυτά τα καινούργια όργανα όπως τις τοπικέ, τοπικές, τις εδαφικές τέλος πάντων επενδύσεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά το σχέδιο κειμένου, να δούμε τι ανάλυση θα κάνετε και να καταλάβουμε τι εργαλεία στην διάθεσή μας και πώς μπορούμε να τα κάνουμε αποτελεσματικά. Και έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Κοινωνικός αποκλεισμό και ρατσισμός. Πρόκειται για δύο κακά τα οποία είναι ριζωμένα μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οπότε Νομίζω ότι είναι όχι απλώς αναγκαίο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια θεσμική συμφωνία μεταξύ τοπικών αρχών, ένωσης, ε, ε κράτων μελών, ώστε να δούμε τι θα γίνει, τι χρηματοδότηση θα γίνει και με ποια από τα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας. Ε, από το 2010 λοιπόν έχουμε το Ταμείο το Κοινωνικό και θα πρέπει να δούμε τι ποσοστό χρηματοδότηση θα γίνει. Και επίσης είχαμε απευθύνει μια σχετική ερώτηση στην ε, Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε δυνατότητες στην πύλη σε αυτούς τους περιθωριακούς και θα δούμε το πώς θα μπορούμε να αποσπάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί εκεί ο κοινωνικός ιστός αλλά η οικονομία και όλα είναι σε πολύ προβληματική κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ε, το Σας ευχαριστώ. Η εκθεσή σας είναι ενδιαφέρουσα. Θα παρακολουθήσω από κοντά την διαδρομή αυτής της έκθεσης και θα προσπαθήσω να βοηθήσω με την εμπειρία που έχω. Πολλά χρόνια έχω κάνει δήμαρχος σε πόλη που είχε αρκετούς τσιγκάνου, οι οποίοι πάρα πολύ συχνά ζουν σε ακίνητα άλλων, οπότε και οι συμπολίτε μας δεν τους ήθελαν εκεί και επίση οι νέοι Ρωμά πολλές φορές ε, στρέφονται στο έγκλημα. Πάντως η κατάσταση τώρα βελτιώθηκε. οι Ρωμά σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να ανελιχθούν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά των Ρωμά και έτσι ε, συνεχίζουμε την πορεία της ένταξής τους. Βελτιώνουμε τις όρους διαβίωσής τους και εξασφαλίζουμε το ότι οι Ρωμά που τώρα γεννώνται θα μπορούν να ζήσουν σαν φυσιολογικοί άνθρωποι στο μέλλον. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να υπάρχουν τέτοιοι αφόρητοι όροι διαβίωση. Θα πρέπει επομένω να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα. Φυσικά και τα δεινά της Ευρώπης δεν έχουν να κάνουν ούτε με τους Ρωμά ούτε με καμία άλλη μειονότητα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το πρόβλημα. Και σας είπα, σύμφωνα με την εμπειρία μου, πρέπει να γίνει η κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων από τη βάση της προκριτικότητας. Δεν θα πρέπει να γυρεύουμε κάποιο κοντόφθαλμο όφελος από τα σχετικά προγράμματα. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι να δώσουμε κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Και φυσικά να δούμε τι αρμοδιότητες ε, έχουν δήμοι, κοινότητες, ε, περιφέρειες και η Ευρώπη επί τη βάση επικουρικότητας. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ τέτοιων ε, λύσεων, όπως προτείνει αυτή η λύση. Χρειάζεται συνύπαρξη. Και εφού θέλουμε συνύπαρξη θα πρέπει να έχουμε διαπραγμάτευση των όρων της κοινή διαβίωσης και της συνύπαρξης με τους Ρωμά. Βεβαίω και είναι κάτι πολύ θετικό το ότι πρόκειται να εκταμιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια χρήματα, οπότε και είναι πιο εύκολο να έχουμε τη διάθεση των πόρων εάν έχουμε εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτά τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Παντού στην Ευρώπη. Μπορεί να αλλάζει κάπως η μορφή τους, να παραλλάσσουν μια χώρα στην άλλη, αλλά Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας και το Κοινοβουλίο γενικό θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση ή στο μέλλον. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σμόλκοβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έσαν με obdržali το dokument. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το εργασία αυτό. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τις ε, παρουσιάσεις σας και είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία που αναφέρονται στη συζήτηση. Και αυτό συνδέεται και με το ζήτημα που συζητήσαμε χθε αργά στην Ολομέλεια. Παρά το γεγονός ότι ακούσαμε και πολύ κριτική. Για καταχρήσεις των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων από τους Ρωμά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τα ζητήματα και τα θέματα κατάχρησης ίσως να αποτελούν πραγματικότητα. Η έκθεση αυτή όμως θα πρέπει να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε μια πραγματική εντύπωση και με ρεαλιστικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Εγώ είμαι από την Ανατολική Σλοβακία και έχουμε πολλούς ε, Ρώμα στην πόλη μου έχω μεγάλη εμπειρία με τα προβλήματα αυτά και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ενεργά να συνεργαστώ. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Allow me to take a... Μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια. Θα τα πω στα βουλγαρικά όμως. Για να σας πω ποια εμπειρία είχα εγώ στα θέματα αυτά και ποια είναι η γνώμη μου. Το uh, Ζήτησα το λόγο για το θέμα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Είναι από τα πιο δύσκολα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και η πατρίδα μου η Βουλγαρία. Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι Βούλγαροι απόδημοι για άλλες χώρες είναι μετανάστες και μερικές φορές οι χώρες υποδοχής έχουν προβλήματα με τους ε, μετανάστες από τη Βουλγαρία. Κάτι που ισχύει και για μετανάστες από άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην ανάγκη ένταξης, κοινωνικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων με έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι μπορούμε να επενδύσουμε για τη βελτίωση των βιωτικών συνθήκων των περιθωριοποιημένων αυτών κοινοτήτων, αλλά αυτό δεν αρκεί και μια τέτοια επένδυση θα πέσει στο κενό αν δεν συνδυαστεί με αλλαγή νοοτροπίας από τις ίδιες τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και δεν δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς ευκαιρία να συμμετέχουν στο κοινωνικό, στο κοινωνικό και οικονομικό βίο και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο με δράσεις ε, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Ας μην το ξεχνούμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Ας το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. γιατί αυτό το στοιχείο της επένδυσης ε, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην παιδεία θα είναι κέριο στην ε, κοινωνική ένταξη αυτών των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Αν επικεντρωθούμε στην παιδεία και στην επαγγελματική κατάρτιση, θα καταφέρουμε να λύσουμε σταδιακά το πρόβλημα της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, να επιλύσουμε το πρόβλημα και όχι να το επιδεινώσουμε αφήνοντα μια κατάσταση να διαιωνίζεται. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να εστιαστούμε μόνο στην κοινότητα των Ρωμά. Και άλλε περιθωρισμένες <coughs> κοινότητε ε, υπάρχουν. κοινότητε ανθρώπων που ε, μεταναστεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και σταδιακά περιθωριοποιούνται γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Αυτά ήθελα να πω ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τώρα να δώσω το λόγο. Δεν βλέπω όμως το όνομά σας παρακαλώ. Ο κύριος Τσβέρ. Μίλα βέρα, ονομάζομαι. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια, γιατί διατέλεσα υπουργό Παιδείας στην πατρίδα μου και το θέμα το Ρωμά ήταν από τις προτεραιότητες του Υπουργείου μου για αρκετό καιρό. Είπατε ότι το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης είναι σημαντικό και θα πρέπει σε αυτό να επικεντρωθούμε για να διευρύνουμε την κοινωνική ένταξη των Ρωμά και να φροντίσουμε και τα παιδιά την ε, έγκαιρη κοινωνικοποίηση τους ε, ξεκινώντας από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τα ε, δημοτικά σχόλια και στην Σλοβενία έχουμε λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη παρουσία των παιδιών κοινοτήτων Ρωμά και στους βρεφονιπιακούς σταθμού και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνήθως μάλιστα έχουμε προβλέψει και το θεσμό του μέντορα Ρωμά που φροντίζει τα παιδιά Ρωμά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, στα δημοτικά, παρακολουθεί την προσέλευσή τους, να είναι τακτική, τους βοηθά στα μαθήματα και το καθεξής. Πιστεύω ότι και με ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κοινωνική ένταξη των Ρωμά στις χώρες μας. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ρωμά δεν είναι η μόνη περιθωριοποιημένη κοινότητα. Υπάρχουν και άλλες αποκλεισμένες κοινότητες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να διευρύνουμε ε, την έκθεση περιλαμβάνοντας και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες. Αυτή θα ήταν η συστασία μου προς την εισηγήτρια. Ωραία. Μια ναι, και δεν βλέπω άλλον ευρωβουλευτή να ζητά το λόγο, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια στιγμή να βάλω τα γυαλιά μου. Έχουμε εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Την κυρία Βιόρενσον και τον κύριο Ντεκέσμακερ από την ε, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και τον κύριο Ορμούς από τη Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ποιο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση απασχόληση είμαι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία ε, Ρένκη για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Καλωσορίζουμε ασφαλώ την πρωτοβουλία αυτή. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικο-οικονομική ε, συνοχή χωρί τη συμπερίληψη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Αυτό είναι σαφέ αντιλαμβανόμαστε τις πολλές προκλήσεις τις οποίες και εντοπίζετε στο έγγραφο εργασίας. Είναι υπερβολικά πολλά στον αριθμό ακόμα, αλλά ελπίζουμε με την θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού της τρέχουσης προγραμματικής περίοδου, διάφορες από τις προκλήσεις που αναφέρατε θα επιληθούν, θα αντιμετωπιστούν. Ο νέος κανονισμός θεωρούμε ότι εισαγάγει κάποια καινούργια μέσα και εργαλεία, τα οποία ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι πολυάριθμες προκλήσεις. Τα ταμεία προορίζονται και προσανατολίζονται πιο πολύ στις πολιτικές, ε, σύμφωνα με τις πολιτικές που αναφέρονται στις εθνικές στρατηγικές για τους Ρωμά. Υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στις επενδύσεις, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις περιθωρισμένες κοινότητες. Και αυτό φυσικά ε, σε συνάρτηση με την ε, διάσταση του mainstreaming. Ο νέο κανονισμό, λοιπόν ενθαρρύνει τι ε, εταιρικέ σχέσει με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και στις ε, σχετικές επιτροπές και επίσης ο κανονισμός δίνει δυνατότητα ενίσχυσης ε, των δυνατοτήτων των ΜΚΟ που συμμετέχουν, για παράδειγμα, για την εκπροσώπηση των Ρωμά. Ελπίζουμε λοιπόν με τους νέους κανονισμούς, με τα νέα εργαλεία τα οποία εισαγάγαμε, κάποιες από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν. Θα προτείναμε ίσως στην έκθεση να γίνει διάκριση μεταξύ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Γιατί όπως σας είπα, ελπίζουμε ότι κάποια από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην προηγούμενη περίοδο θα έχουν αντιμετωπιστεί για την τρέχουσα περίοδο. Τέλος, θα ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε εδώ σε καθεστώς ε, κοινή διαχείρισης και θέλουμε φυσικά να συμμετέχουν, να όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ευχαριστώ πολύ. Μία πρακτική Ερώτηση, μπορείτε να μα ενημερώσετε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά σα. Θα θέλαμε εμεί η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή να μάθουμε για να δούμε πώ θα γίνει για να ολοκληρωθεί η διαδρομή τη έκθεση. Καλώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρέντικε, θα θέλατε να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα σχολιάσατε. Να ξεκινήσουμε με το πρακτικότερο θέμα. Έχουμε το σχέδιο κειμένου στην Επιτροπή 4 και 5 Μαΐου. Οπότε αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Και στη συνέχεια πρόκειται να ψηφίσουμε την κατάσταση λίγο πριν τις ε, διακοπές και θα κατέβει στην Ολομήνια του Σεπτεμβρίου. Πολλά και αξιόλογα ε, ακούσαμε και όλα αυτά τα, τα έχουμε υπόψη μας ε, τώρα εν ώψη του σχέδιου κειμένου το οποίο θα συντάξουμε. Επίσης είχαμε το θέμα του ορισμού το οποίο ανέκυψε σε πολλές ε, παρεμβάσεις και σας διευκρινίζω ότι στις επαφές και συζητήσεις μας δεν ζήτησαμε μόνο με εκπροσώπους και φορείς των Ρωμά αλλά μιλήσαμε αρκετά και με άλλους εμπλεκομένους κοινωνικές πλατφόρμες, την ε, το Solida κλπ. Και ε, βεβαίω αυτά που μάθαμε από τη συζήτηση είναι ότι έχουμε και άλλες μειονότητες περιθωριοποιημένες, αλλά η Ρώμα είναι πιο μεγάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές είναι εκείνοι οι οποίοι υφίστανται περισσότερο τον αποκλεισμό και πιο έντονα τις δυσμενείς διακρίσεις. Αυτό θέλουμε να ξεκαθαριστεί ε, και στο έγγραφο εργασία, αλλά και στην έκθεση. Και θα έχουμε τέτοιου είδου προσέγγιση να γίνει. Τώρα, κι άλλα. Ε, ακούσαμε που τα οποία ακόμη τα ερευνούμε. Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλου όσον αφορά την άλλη των δεδομένων. Δηλαδή, πώ την τελευταία χρονοδοτική περίοδο έγινε η δαπάνηση των πόρων. Και τι θα γίνει με τη νέα χρηματοδοτική περίοδο, τι θα γίνει με τον νέο κανονισμό, ο οποίο υποτίθεται ότι θα επιλύσει κάποια από τα προβλήματα αυτά τα οποία αναφέρονται στο έγγραφο εργασία. Βλέπουμε και τι εταιρικέ συμφωνίε, βλέπουμε αυτά τα επιχειρησιακά λειτουργικά προγράμματα και θα δούμε τι θα γίνει τη νέα περίοδο, γιατί τα προβλήματα ακόμα υπάρχουν. Οπότε αυτό θα πρέπει να τα συζητήσουμε και άλλο. δεν είναι μόνο θέμα καινούργιου κανονισμού που θα λύσει ξαφνικά όλα τα προβλήματα. Η ε, Κύριε Ντεμάτη, είπε το πώς θα συνδυάσουμε την προσπάθεια αυτή με άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Και μία από τις ιδέες είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Και να δούμε πώς θα καλύψουμε μέσω αυτού και τις περιθωρισμένες κοινότητες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρατε κύριε όσον αφορά την ε, απασχόληση. Γι' αυτό να δούμε πώς θα γίνει ο συνδυασμός και πώς θα μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν τις διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Γυναικών ε, πρόκειται να είναι συναρμόδια και θα φτιάξει μια έκθεση. Είναι σημαντικό πάντως. Επίσης, και το Κοινωνικό Ταμείο έχει σχέση με το αντικείμενό μας. Επίσης η Επιτροπή Απασχόλησης θα συντάξει κάποια έκθεση. Θα δούμε τώρα την εκπαιδευτική διάσταση. Γιατί έχουμε αυτούς τέσσερις τομείς. Εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγαση. Θα πρέπει να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη άποψη και να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολιτική συνοχή και όλα αυτά να τα συγκεράσουμε και έτσι να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών στην Ευρώπη. Και να του εμπλέξουμε σε όλε τι φάσει τη ε, συζήτηση και προβληματική. Ε, αυτό θα είναι βήμα πρόοδου. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όσο λέω. Ε. Μιλούμε για τους περιθωριοποιημένους αλλά θα πρέπει να είναι περιθωρημένη και η συζήτηση και η θέση τη συζήτηση στην ημέση διάταξη. Συμφωνώ. Και με την Επιτροπή Ασχόληση και με την Επιτροπή των Γυναικών πρόκειται όλα αυτά να τα βάλουμε στη, σε κορυφαία θέση ε, στο θεματολόγιο του Κοινοβουλίου και να δούμε τι θα γίνει. Να έχουμε και τη Διεθνή ημέρα για τους Ρωμά. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους, να συνεργαστούμε ψηλή προτεραιότητα και έτσι να λύσουμε το πρόβλημα της ε, ε, περιθωριοποίησης ε, για όλες τις μειονότητες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα. Συνεχίζουμε με το σημείο 14. Συζήτηση και εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Ο συντάκτης της γνωμοδότησής μας είναι ο κύριος Ανδρέα Κοτσολίνο. Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού. Εμείς θα συντάξουμε γνωμοδότηση, την οποία θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Μαΐου. Η προθεσμία για τις τροπολογίες θα λήξει στις 12 το μεσημέρι, ημέρα Δευτέρα 13 Απριλίου, ώστε να είμαστε έτοιμοι για την, να ψηφίσουμε το Μάιο. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι, έχει σημαντικό ρόλο στην πρόθεση της ε, ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και πολλές ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, πρωταγωνιστούν στο θέμα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε και ανακοίνωση με θέμα την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας θα συντάξει έκθεση επί της ουσίας και εμείς γνωμοδότηση. Και αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση γιατί η πολιτική συνοχή είναι σημαντική πηγή χρηματοδότησης ε, σχεδίων υποδομών για τον πολιτισμό. Και μάλιστα στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ε, περί 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν σε πολιτιστικά προγράμματα, 15 πλάσιο από τον ε, συνολικό προϋπολογισμό για την παιδεία στην προηγούμενη περίοδο. Αυτέ ήταν οι επενδύσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξη. Κύριε Κοτσολίνα, έχετε το λόγο. Θα είμαι σύντομα και πρόκειται για μια πολιτική η οποία συμβάλλει περισσότερο όσον αφορά αυτές τις, τις, αυτούς τους πόρους γιατί πρόκειται για έναν τομέα εδώ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, ζωτικότητα και από πλευρά ευρωπαϊκή ταυτότητας. Αλλά έχει σημασία και οικονομική όσον αφορά την παραγωγή πλούτου και απασχόλησης. Οπότε μιλούμε τώρα για πάρα πολλές ΜΜΕ ε, οι οποίες είναι και καινοτόμε και έτσι καθορίζεται ε, το τι γίνεται και με τι τις ροές του τουρισμού. Ε, οπότε θα πρέπει να δούμε με τους σπόρους. Δεν τα διαβαίνω τόσο γρήγορα γιατί ακριβώ αυτή η πολιτική περιλαμβάνει πολλές ποικίλε δραστηριότητε. Άρα εμείς θα γνωμοδοτούμε, η Επιτροπή Πολιτισμού είναι κυρίως αρμοδία και εμείς θα επισημαίνουμε από πλευράς μας τρία τεινά. Πρώτα-πρώτα τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιφραγών προγραμμάτων για την χρήση των πόρων. Έχουμε αυτή την πολιτική των μεγάλων προγραμμάτων, οπότε και είναι πάρα πολύ σημαντικό τι είδους επιλογές θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα συσχετίσει με την υπόθεση αυτή αυτά τα 5 εκατομμύρια ε, για, τις, ε, για, τα, για τα προγράμματα της UNESCO και τα άλλα 10 εκατομμύρια που επίσης που προβλέπονται. Οπότε, πρόκειται τους τόπους αναγνωρισμένους από την UNESCO. Είναι σημαντικές αυτές οι δράσεις της Επιτροπής, είναι θέμα που το συζητούν παντού. Ε, υπήρχε αυτό το μεγάλο έργο της Πομπίας και εδώ ε, αναφέρονται αυτές οι επενδύσεις, τα 10 και τα 5 εκατομμύρια. Θεωρώ ότι αυτή η προοικοδότηση δεν αρκεί και θα πρέπει τελικά να διατεθούν γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια παρατήρηση είναι αυτό το οποίο το συζητήσαμε πρόσφατα πως δηλαδή αυτή η πολιτική που έχει σχέση με την πολιτική της συνοχής πως θα συσχετιστεί με το πλάνο Juncker πώς θα έχουμε τη συμμετοχή, την εμπλοκή, την επιλογή των ε, projects, πώς θα εμπλακούν εδώ οι ιδιώτες, γιατί πρόκειται εδώ για πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει πάρα πολλής χώρος εδώ και ευκαιρία για την ιδιωτική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να συνοδεύσει ε, τη, τους πόρους τους κοινοτικούς. Τρίτη παρατήρηση έχουν πάρα πολύ στενή σχέση αυτές όλες οι πολιτικέ. Α πούμε το Horizon 2020 με αυτήν ε, τον νέο προγραμματισμό για τη διάθεση των πόρων 2014-2020. Όμως βέβαια οι προσεγγίσει είναι διαφορετικέ. Δύο διαφορετικέ προσεγγίσει υπάρχουν επομένω. Αυτά ήθελα να σα πω και βέβαια θα λάβω υπόψη και έχουν να πούν στη συζήτηση οι άλλοι συνάδελφοι προ, πρόθυμο σήμερα να καλύψω όλες τις προτάσεις τους αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά θέματα και θα πρέπει ε, να συμβάλλουμε με αυτά τα στοιχεία που σας είπα στο έργο της ε, κυρίως αρμόδας Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε τον κύριο Σβέρ που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Κοτσολίνο που ε, μας παρουσίασε το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συνολική προσέγγιση. Είμαι μέλος και της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Αναπληρωτής ε, εδώ. Θα ψηφίσω λοιπόν και για το ψήφισμα. Επιτρέψτε μου όμω να κάνω κάποιε σύντομες παρατηρήσει. Θα μπορούσε να έχει επιδείξει λίγο παραπάνω φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προετοίμασε αυτή την πρόταση. Ακόμα και στον τίτλο τον ίδιο. Αν δεν μιλάει για ολοκληρωμένη προσέγγιση, το οποίο ακούγεται λίγο διεκπαιρετικό, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις οικονομικές ε, δυνατότητες αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν έχει μόνο δυναμικό οικονομικό, αλλά καθορίζει και την ίδια μας την ε, ταυτότητα. Ο κόσμος ε, έχει διάφορα είδη ταυτότητας ευρωπαϊκό εθνικό, σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο, σε πολιτιστικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Να μην υποτιμούμε και την οικονομική πτυχή σε ό,τι αφορά δηλαδή και τις ε, θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει επίσης και ο παράγοντας της συνοχής. Υπάρχουν ε, πραγματικά πολιτιστικά μνημεία ύψης της σημασία σε περιοχές που δεν αναπτύσσονται ε, απαραίτητα όσο θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν αυτή η πτυχή της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτρέπει στην Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική. Δεν είμαστε οικονομικοί φορείς ε, υψηλής, αν θέλετε κορυφαίοι ή στρατιωτικά δεν είμαστε οι πιο δυνατοί. Από γεωγραφικής άποψης δεν είμαστε, από δημογραφικής άποψης επίσης δεν είμαστε οι γίγαντες, αλλά σε επίπεδο πολιτιστικό έχουμε μεγάλη κληρονομιά να επιδείξουμε, για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην σε τη παραγωγή ταινιών είμαστε σε δεύτερη θέση στην ε, παραγωγή βιβλίων, στον αθλητισμό. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ευρώπη κερδίζει τα πιο πολλά βραβεία και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια έκφανση της καλής ποιότητας ζωής που έχουμε στην Ευρώπη και το, η οποία θα πρέπει να προστατεύεται στο μέλλον, να προσδεθεί στο μέλλον. Αυτά για να σας πω ότι δεν πρόκειται μόνο για ηλική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για το είδος ζωής που διάγουμε. Έχουμε την ψηφιοποίηση ασφαλώς της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό χρειάζεται και πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση. Να αναφέρουμε επίσης ε, το δυναμικό του επενδυτικού προγράμματος του Juncker προς την κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι το ανέφερε και ο ίδιος ο εισηγητής. Χαίρομαι λοιπόν που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Είναι ως στη φύση του. Δύο επιτροπές εξετάζουν τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ιάκοφτσιτς, έχετε το λόγο. <coughs> Οι μελλοντολόγοι <coughs> λένε ότι η Αμερική θα γίνει ε, εμπορικό κέντρο, η Ασία εργοστάσιο παραγωγής, η Αφρική ε, θέρετρο και η Ευρώπη μουσείο. Τι να σας πω, μελλοντολόγια τα λένε αυτά. Πάντως ε, είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στη βελτίωση του σχεδίου γνωμοδότηση, ιδιαίτερα στο τμήμα που αφορά την ύψη της αξίας πολιτιστική μας κληρονομιά, που είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί η συγκέντρωση πολιτιστικών μνημείων της UNESCO στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι τεράστια. Αλλά δεν μιλούμε μόνο για υλική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για άειλη πολιτιστική κληρονομιά, που επίσης ε, είναι εξαιρετικής αξίας καλή πρωτοβουλία. Θα συμβάλλουμε και εμείς στην γνωμοδότηση. Ας θύμα μακρηγορήσω. Θα βοηθήσουμε και θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. κυρία Ρέντκε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης και ε, εμεί ε, συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά στην Ευρώπη και διαβάζοντας το κείμενο σκέφτηκα ότι αυτό που θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, είναι να μην επικεντρωθούμε μόνο σε μεγαλεπίβολα πολιτιστικά σχέδια και προγράμματα, αλλά να δείξουμε ότι οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες ο και ο τομέας της δημιουργικότητας και της ευρηματικότητας ε, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό θετικό ρόλο στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί είναι τομές ε, οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλουν στην οικονομία. Και από αυτήν την άποψη θα πρέπει να στηρίξουμε πιο τοπικά, περιφερειακά προγράμματα πολιτιστικά μικρής κλίμακος και όχι μόνο τα μεγάλα επίβολα, γιατί ακριβώς τέτοια μικρή κλίμακα ε, τοπική εμβέλεια προγράμματα μπορούν να τονώσουν την ανάπτυξη και ταυτόχρονα να διαφυλάξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Λέμε και στο έγγραφο ότι οι επενδύσει στην πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντικέ. Και χάρη στην γνωμοδότηση αυτή και στην έκθεση τη Αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την φόρα που πήραμε και να διατρανώσουμε την πρότασή μας να αποτελέσουν οι επενδύσεις στα πολιτιστικά θέματα προτεραιότητα της Ευρώπης. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Κοτσολίνο, για την νομοδότησή σας. Να σου πω πρώτα τα καλά βουλό και μετά τα στραβά. Εδώ μιλούμε για τη δυνατότητα που έχουν να αναδειχθούν αυτού του είδους τα έργα για, για τον πολιτισμό, αλλά για την έρευνα και τις ΜΜΕ. Και εδώ πέρα μας τονίζεται πώς μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους ε, projects τα οποία είναι δυνατόν να συνδεθούν με την αξιοποίηση της ε, πολιτικής οικονομίας. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, της επικουρικότητας και παράδειγμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το ότι έχουμε αυτή την πλατφόρμα Valor και ε, μέχρι σήμερα έχει ε, δημιουργηθεί μόνο η και για το Creative Europe. Άρα να κάτσουμε και να δούμε ε, τι θα υπαχθεί εδώ. Δεν είναι όλη η υπόθεση όμως εδώ τα μεγάλα έργα. Και επίσης αναφέρατε εδώ πέρα σαν παράδειγμα το έργο στην Πομπία, αλλά αυτό δεν είναι τόσο εύστοχο νομίζω γιατί και η κυρία Κρέτου, η Επίτροπος μα είπε ότι υπάρχει κίνδυνο να μην εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα. Λέτε εδώ για 150 εκατομμύρια ευρώ ε, και 35 από, την, από την, τα κράτη, αλλά είπαμε για 47 εργοτάξια, αλλά δεν ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα πρέπει να τονιστεί πιο πολύ η σημασία του πολιτισμού για την ε, ανάπτυξη. Κυρία Γουόρ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Γιατί θα πρέπει να προσέξουμε να μην μιλήσουμε για το παρελθόν, να μιλήσουμε για το μέλλον και να έχουμε πάντα το μυαλό μας το παρόν. Νομίζω ότι λείπει ίσως κάτι. Η διάσταση του πώς το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει για ένα καλύτερο μέλλον. Και έχουμε πολλά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη για που θα μας θυμίζουν τα λιγότερα έντοξα κομμάτια της ιστορίας μας. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη που είναι σε πραγματικό κίνδυνο εξτρεμιστικών δυνάμενο να εντοπίσει και να συμπεριλάβει και να προσπαθήσει να επιστήσει την προσοχή σε κάποια μνημεία συνείδησης που υπάρχουν όχι μόνο μέρη όπως το Auschwitz, αλλά και άλλα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, όταν παραβρέθηκα στην Βουδαπέστη πριν από κάποια χρόνια, επισκέφτηκα ένα πολύ μικρό μουσείο όπου οι μυστικές υπηρεσίες βασάνιζαν πολίτες. Ήταν πραγματικά τεράστιος ο αντίκτυπος που μου έκανε. Ήταν ένα μικρό καθημερινό κτίριο, το οποίο όμως με επηρέασε τεράστια. Θεωρώ ότι έχουμε καθήκον λοιπόν να διαφυλάξουμε και αυτές τις πλευρές της ιστορίας για να θυμόμαστε γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, ο κ. Βανίσερο. Συντομία. Η κυρία τη Σκιώδης από την ομάδα μας δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά μου άφησε κάποιες σημειώσεις Κάντε και στη βέβαια κάποια σχόλια. Είναι πραγματικά μεγάλη και πλούσια η κλημορφία μας στην κατάρτιση των πολιτικών μας ε, σήμερα, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μιλάμε για ευθυή e e εξειδίκευση. Μία μέθοδο όπου μαρετούμε διάφορες υποθέσεις και πτυχές ενός ζητήματος για να μάθουμε καλύτερα το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις λειτουργικότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είτε πρόκειται για κτίρια, είτε πρόκειται για είδος ζωής και πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Για το πώς μπορούμε δηλαδή αυτά τα πολυάριθμα μνημεία που έχουμε να τα αξιοποιήσουμε. Που πρέπει να τα πληρώνουμε, γιατί είναι τόσο πολυάριθμα για παράδειγμα τα μνημεία της Ιταλίας που σκεφτείτε τι ποσά δαπανώνται ή πρέπει να δαπανηθούν για να τα διατηρούν αυτά, να τα συντηρούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε από αυτά με σύγχρονο τρόπο, πώς μπορούμε να τα προαγάγουμε στον τουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο. Πώς μπορούμε λοιπόν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να συνδέσουμε τα μνημεία αυτά με τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Με μία οικονομία, με βάση τη γνώση ευθύης εξειδίκευση και εδώ. Επίσης είναι καλό ότι υπάρχει αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μπορούν να αξιοποιηθούν και να δημιουργηθούν διάφορα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, συνοχής, θαλάσσια, τα, ταμεία θαλάσσιας ανάπτυξης για τις παράκτιες ε, περιοχές για να προσελκύσουμε νέο τουρισμό, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Επίση, πώς παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την όλη διαδικασία αυτή, είναι τόσο ανοιχτό το θέμα αυτό. Πιστεύω, για παράδειγμα, για να είμαι ειλικρινής, ότι ο καινούργιος κανονισμός είναι πολύ πιο περιοριστικός. Γιατί αν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία της προηγούμενης ε, προγραμματικής περίοδου, δεν έχουμε καθόλου καμία ιδέα για το κατά πόσο θα, πώς θα εξελιχθούν τα στοιχεία αυτά για τα λειτουργικά προγράμματα. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να μας ενημερώνει. Το γεγονός των 5 εκατομμυρίων ευρώ αν συνδυαστούν για διάφορες χρηματοδοτήσεις, τα διάφορα κοντήλια. τα 5 εκατομμύρια δεν είναι πολλά. Ζητούμε λοιπόν και ευελιξία. Αυτά λοιπόν από δική μα πλευρά και πήρε το λόγο και ο κύριο Βέτ. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί, παρακαλώ. Επειδή είμαι και μέρο τη επιτροπή, ε, επιτρέψτε μου να ξαναλάβω το λόγο και πάλι στα βουλγαρικά. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Η, η γνωμοδότηση το κυρίου Κοτσολίνο είναι πολύ σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη σε πολλά κρατημέλη. Και η πρακτική χρηματοδότησης ε, σχεδίων που προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά μας επιτρέπει να μετατρέψουμε την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό αγαθό και να στηρίξουμε και την τοπική οικονομία. και άρα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των περιφερειών. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε και καλή εξειδίκευση των μεμονωμένων περιφερειών. Και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε στρατηγικές για να προβάλλουμε την πολιτιστική κληρονομιά και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Επίσης, να προσφέρουμε κατάλληλες υπηρεσίες ε, για την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο σε μεγάλα πολιτιστικά προγράμματα, γιατί έχουμε πολλά μικρά προγράμματα που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση για να διεκπαιρεωθούν. Μερικές φορές μερικά προγράμματα σταματά στη μέση επειδή στερεύουν τα κονδύλια. Είναι κρίμα να μην μπορεί η πολιτική συνοχή να χρηματοδοτεί μέχρι τέλους ένα πρόγραμμα. Και μάλιστα στη Βουλγαρία προβλέπουμε ειδική πρόσβαση στα επιχειρησιακά προγράμματα μέσω της προτεραιότητας που έχουμε για την ανάπτυξη των ε, πολιτιστικών μνημείων. Και των ε, αξιοθεάτων. Έχουμε έτσι πολλά αξιοθέατα στη Βουλγαρία και πολλά ε, μέρη ανεπτυγμένα τουριστικά με πολιτιστική κληρονομιά και έτσι με την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών προς τους τουρίστες αναπτύσσεται και η τοπική οικονομία. Σημαντικό επίτευγμα της Βουλγαρίας στον τομέα αυτό. Φυσικά χρειάζονται και επίβολα προγράμματα σαν αυτό της Πομπίας, γιατί η Πομπία είναι μοναδικό μνημείο στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει κάθε περιφέρεια να εκπονήσει τη δική της στρατηγική και το δικό της στρατηγικό όραμα για να χρηματοδοτήσει και μικρότερες εμβέλειες σχέδια που θα προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη. Αν θέλει άλλος κανείς το λόγο, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στους εκπροσώπους. Έχουμε ε, εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού και από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ποιος θέλει πρώτα στο λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ε, είμαι επικεφαλής της ομάδας ε, ε, περιφερειακής αποδοτικότητας. Να ξεκινήσω λοιπόν με το βασικό και το πιο εύκολο τμήμα της παρέμβασης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε τα πιο πολλά όπως ακούσαμε εδώ σήμερα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά τονίζει τη σημασία της πολιτισμικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συζητήσεις για το νέο προγραμματικά έγγραφα υπογραμμίζει τη σημασία μιας ενοποιημένης, ολοκληρωμένης προσέγγισης στην πολιτιστική κληρονομιά. Σε διάφορους βαθμούς βλέπουμε στα κρατημέλη όντως ότι και αυτά δίνουν μεγάλη σημασία στην πολιτιστική κληρονομιά. Ένα παράδειγμα στις αρχές του μήνα το νέο λειτουργικό σχέδιο για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη της Ιταλίας εγκρίθηκε με 500 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020, καλύπτοντας πέντε περιοχές περιφέρειες της ε, Νότιας Ιταλίας. Άρα η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμο και σημαντικό κομμάτι της ε, πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Να στραφούμε στα πιο δύσκολα τώρα. Τμήματα της συζήτηση, ε, όπως έθιξαν και κάποιοι βουλευτές, το θέμα του κατοφλιού των 5 ή 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον πολιτισμό και τις κριτικές υποδομές για τον τουρισμό. Αυτό προέρχεται κατευθείαν από τον κανονισμό για την περιφερειακή ανάπτυξη όπου ορίζονται τα διάφορα είδη υποδομών τα οποία μπορεί να υποστηριχθούν από το Ταμείο μια μεγάλη λίστα, ενέργεια, περιβάλλον, ε, επιχειρήσεις, εκπαίδευση και μετά αλλάζει η διατύπωση σε ό,τι αφορά τον, την υποδομή για τον τουρισμό γιατί περιγράφεται ως μικρής κλίμακας και είναι σημαντικό αυτό ως επίθετο γιατί αυτό τροποποιεί την κλίμακα των έργων που μπορούν να υποστηριχθούν. Μικρής κλίμακας μπορεί να περιλαμβάνονται μόνο μπορεί να αφορά, το μικρής κλίμακας μπορεί να αφορά μόνο την οικονομική πτυχή. Η σημασία της υποστήριξης ε, των υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς που μάλλον η πολιτιστική υποδομή είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν περιλαμβάνει όλη την πολιτιστική κληρονομιά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να επιδείξουμε όσο πιο μεγάλη ευελιξία γίνεται, σεβόμενη παρόλα αυτά την ακριβή του κανονισμού. Το όριο των 5 εκατομμυρίων από πλευρά μα θεωρούμε ότι αποτελεί πολύ γενναιόδορη και ευρεία ερμηνεία του επιθέτου μικρής κλίμακας του προσδιορισμού μικρής κλίμακας. Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλους κανονισμούς και διδάξεις, το μικρής κλίμακας συνεπάγεται έργα 250.000. Τα 5 εκατομμύρια λοιπόν είναι πολύ γενναιότερη ερμηνεία. Σε συνδυασμό με αυτό μιλάμε για επενδύσεις ε, σε υποδομές ε, μικρές υποδομές ε, μικρής ε, εξειδίκευσης. Και η Πομπία ε, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε την προσέγγιση ότι μιλάμε σε μεμονωμένα ότι μιλάμε για μεμονωμένα τμήματα υποδομών. Άρα για μεμονωμένα τμήματα υποδομών σεβόμαστε το όριο, αλλά αυτά μπορούν να αποτελούν μέρος ενός αθροίσματος. Και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει για το μνημείο της Πομπίας. Όπως σας είπα, εξαρτήσαμε στο βαθμό του δυνατού την ευελιξία μας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και όρια από πλευρά ερμηνεία. Αυτή είναι η προσέγγιση την οποία ακολουθήσαμε. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα τα κράτη-μέλη ήταν ευχαριστημένα με την προσέγγιση αυτή, αλλά έγινε αποδεκτή αυτή η προσέγγιση, αυτά τα όρια. Και νομίζω ότι αυτό που είπαμε στα κράτη-μέλη είναι ότι έχουμε ήδη διάφορες ε, αμφιλεγόμενες περιπτώσεις και θα πρέπει να τα συζητούμε πάντα αυτά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των προτέρων για να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εμείς ευχαριστούμε, Λεπρόεδρος. Τελειάλος το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στο ζωηρό ενδιαφέρον σα την πολιτιστική κληρονομιά και πέρυσι, όταν δημοσιεύσαμε την ανακοίνωσή μα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, το κάναμε γιατί είχαμε επίγνωση το συνεπειών που έχει αυτή στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ταυτότητα των πολιτών, στην ευρωπαϊκή ταυτότητα γενικώ. Και επίση επηρεάζεται η περιφερειακή πολιτική, ή ε, μάλλον η πολιτιστική κληρονομιά από άλλε πολιτικέ. Και με την, με την πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη θα στηρίξουμε ιδιαίτερα την πολιτιστική κληρονομιά. Ήδη λοιπόν έχουμε αρχίσει το έργο που αναγγέλαμε στην ε, ανακοίνωση ολοκληρωμένης προσέγγιση. Ήδη έχουμε συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, ε, συλλέγουμε τις βέλτιστες πρακτικές για τους καλύτερους τρόπους συμμετοχικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Και του χρόνου θα ολοκληρώσουμε τη συλλογή των βέλτιστων πρακτικών και θα δημοσιεύσουμε τα πορίσματα αυτής της μελέτης. Σας ευχαριστώ. Έχω και άτυπα κάποιες ερωτήσεις. Τα 5 εκατομμύρια είναι η συμβολή του Ταμείου, η συνεισφορά του Ταμείου, θα είναι το σύνολο του προγράμματος. Πολλές λεπτομέρειες έχουμε να λύσουμε εδώ για, το, για τη χρηματοδότηση μικρής εμβέλειας. Δεν λέω ότι θα λάβουμε και απαντήσεις, απλώς στροφή για περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ και ξαναδείτε το λόγο στον εισηγητή σας, διδάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Κοτσολίνο. Λίγες σκέψεις. Στη συζήτηση είχαμε αυτό το θέμα της ερμηνείας της ευέλικτης σημεί του άρθρου 3. Και ποια είναι η σημασία των 5 εκατομμυρίων για ένα έργο που μπορεί να έχει σχέση με επενδύσεις. Οπότε θα μπορούσαμε να φέρουμε πέραν της φομπίας και πολλά άλλα μεγάλα έργα. Να δούμε το θέμα πώς θα μπορέσει να αναδειχθεί η αξία του κάθε τόπου που είναι ο καθένας μοναδικός. Πολλέ φορέ δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί δεν τα τώρα. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Και για ένα άλλο λόγο το λέω. Ξέρω πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Και βέβαια αυτός ο τόπος ανήκει στην Ιταλία Και επίσης ε, τι γίνεται με τις δικαστικές αυτό είναι άλλο θέμα. Και η χρήση των κοινωτικών πόρων επίσης είναι ένα θέμα. Προς το παρόν υπάρχει εδώ υποαπορρόφηση, άρα θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει η διαχείριση όταν έχουμε κάποιες, ε, ε, κάποιους πόρους για κάποιο έργο Μιλούμε για κάποιες ανασκαφές που αφορούν 23 εκτάρια. Άρα ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά. Καθίστε να φανταστείτε τι μπορεί να γίνει ακόμα στην Πομπία. Τέλος πάντων, μην συζητάμε για αυτό. Ναι, χρειάζεται ευελιξία και προς τα πάνω. Λοιπόν, δεν διακυβεύεται τώρα η σημασία της πομπίας, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει πιο καλή διαχείριση και έλεγχος και της χρηματοδότησης των 6 δις, τα οποία ε, διατέθηκαν στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Επίσης πρέπει να σας επισημάνω ότι το θέμα εδώ δεν είναι οικονομικό. Είναι θέμα ταυτότητας, κύρους, ιστορίας και ζωτικότητας της Ευρώπης και γι' αυτό και τα τονίζουμε. Τα ψηφιακά, όλα αυτά τονίζονται στην έκθεση. βεβαίω και τις προτάσεις θα προσπαθήσω να τις καλύψω, να συνεργαστούμε και τελικά να υπάρξει μια έκθεση ευρεία συνένεση στην Επιτροπή μας. Κύριε Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ και σας υπενθυμίζω συνάδελφοι ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 13 Απριλίου το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στις 5 Μαΐου. Το επόμενο θέμα σήμερα στη διάταξη είναι η έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Σήμερα το πρωί συνεδριάσαμε και σας εστάλησαν οι αποφάσεις με email. Έχετε κάποια ένσταση? Όχι από ό,τι βλέπω. Επομένως εγκρίνονται αυτές οι αποφάσεις. Κάτι άλλο για τα διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Και το τελευταίο θέμα σήμερα στη διαταξή σας είναι ότι η επόμενη συνεδρίασή μας πρόκειται να γίνει τον Μάιο. 4 Μαΐου. Από τις 3 μέχρι τις 6 και μισή. Και στις 5 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Τον τελευταίο στοιχείο από Να αναφέρω ευχαριστούμε τους ε, διερμηνείς για το έργο του σήμερα και επίση να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους αλλά και προσκεκλημένου πέρα στη συνεδρίαση.